Καλημέρα σε όλους σας όσοι είστε παρόντες εν πάση περιπτώσει. Θα ξεκινήσουμε έστω και αν δεν έχουμε μεγάλη ε, ε, παρουσία των μελών. Θα ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλές εργασίες, έχουμε εισηγητές οι οποίοι βεβαίως ε, έχουν και άλλες δεσμεύσεις και επομένως θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάποιες ανακοινώσεις εξ ονόματος της Προέδρου Σαρτόρη. Η πρώτη είναι ότι η, συνεδρίαση της κοινής, η κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής για ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά ε, τον ορίζοντα 2030 θα λάβει χώρα αύριο, αύριο στις 3 το απόγευμα. Από τις 3 μέχρι τις 6 προβλέπεται Έχουμε αυτή την αλλαγή λοιπόν. Μια άλλη αλλαγή αφορά το σημείο 7, δηλαδή την παρουσίαση εξ ονόματος της Επιτροπής της ε, δέσμης ε, της Επιτρόπου Κρός για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ήταν ε, γεγραμμένο το σημείο αυτό ε, σήμερα, θα γίνει σήμερα, αλλά όχι σαν σημείο 7, αλλά σαν σημείο 3 μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το σχέδιο δράσης για την Χαλιβουργία. Επίσης, το σημείο της συναδέλφου Φόρντ ε, ε, θα αλλάξει θέση με το θέμα της κυρίας Ουλβσκοκ, τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις εγκατάστασης εφιών δικτύων. Δεν φορά ούτως ή άλλως <clears throat> το πρόγραμμα του της πρωινής συνεδρίασης. Επίσης, η επόμενη συνεδρίαση Ήτρε θα λάβει χώρα στις 17 Οκτωβρίου, 7 με 9.30, στο Στρασβούργο λοιπόν. Είναι μία από τις έκτακτες αυτές συνεδριάσεις που κάνουμε στο Στρασβούργο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον συνάδελφο Γκιούρκο που είναι εισηγητής έτσι ώστε να παρουσιάσει το σχέδιο βράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλιβουργία στην Ευρώπη. Κύριε συνάδελφε παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω ε, που είναι δυνατόν η Ήτρε να εξετάσει την ε, σημερινή κατάσταση στην ε, Χαλιβουργία και τις προοπτικές μέσω έκθεσης πρωτοβουλίας. Είναι βιομηχανία κλειδί που μας δίνει σημαντικές πρώτες ύλες για άλλες μεταπητικές βιομηχανίες, για τον ηλεκτρονικό τομέα, τον τεχνολογικό τομέα, την αυτοκινητό βιομηχανία Η σημασία της ε, χαλιβουργίας ε, συνδέεται με την σημασία που είχε για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πρώτο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Και αυτό που έκαναν οι ιδρυτικοί πατέρες ε, της Ευρώπης ήταν να επιχειρήσουν να συντονίσουν τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό. Η οικονομική ανάπτυξη και η μακροπρόθεσμη προστασία του περιβάλλοντος θα ήταν αδιανόητη χωρίς την ενεργό συμμετοχή και συμβολή της χαλιβουργίας. Οι καινοτόμες διαδικασίες μας επιτρέπουν να έχουμε αποτελεσματική και βιώσιμη εκμετάλλευση, για παράδειγμα για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις ανεμογεννήτριες έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης χωρίς να χάνουμε ε, την ποιότητα των προϊόντων. Γι' αυτό μας βοηθάει να διατηρήσουμε τους πόρους για τις μελλοντικές γενιές. Η Ευρώπη έχει το 11% της παγκόσμιας ε, παραγωγής χαλιβουργικών προϊόντων και πάνω από 500 χαλιβουργία υπάρχουν στα 23 κράτη-μέλη της Ευρώπης που δίνουν άμεση απασχόληση σε 363.000 ε, εργαζόμενους. Και ενώ αυξάνεται συνέχεια παγκοσμίω η παραγωγή χαλιβουργικών προϊόντων λόγω της αύξηση της Κίνας, η ε, ευρωπαϊκή χαλιβουργία είναι σε πολύ αδύναμο σημείο, διότι είναι μειωμένη η απέτηση για τέτοια προϊόντα στην Ευρώπη. Για να τονίσουμε επίσης ότι από το 2009 υπάρχει κρίση στη χαλιβουργία και δεν υπάρχει ε, ανάπτυξη ε, μόνιμη σε κανένα τέτοιο τομέα και έχουμε και κάποια συγκριτικά μειονεκτήματα λόγω της κρατικές, ε, των κρατικών επιδοτήσεων αντισώμενες χώρες και των υψηλών τιμών ενέργειας. Και γι' αυτό ανησυχούμε ιδιαίτερα, διότι η κρίση σημαίνει και η παρατηνόμενη κρίση σημαίνει ότι έχουν μειώσει πάρα πολύ το δυναμικό παραγωγή στην Ευρώπη οι χαλιβουργίες ή και έχουν κλείσει χαλιβουργία, κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει 40.000 θέσει εργασία. Για οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού λόγου και για την ασφάλεια τη ε, ε, προμήθειας έχει μεγάλη σημασία η Ευρώπη να συνεχίσει να είναι βασικός χαλιβουργός και στο μέλλον. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε το 2012 μια ανακοίνωση για τα χαλιβουργία για να αναπτύξει την παραγωγή μας στον τομέα αυτό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση για το 2013, το πρόγραμμα δράση για τη χαλιβουργία έχει μεγάλη σχέση με το θέμα αυτό. Πριν εξετάσουμε τις ε, κύριες ε, προκλήσεις στον τομέα αυτό, θα πρέπει να εξετάσουμε τους παράγοντες που παίζουν ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής χαλιβουργίας. Ε, τέσσερα σημεία συνοψίζουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χαλιβουργία στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα, υψηλό κόστος της ενέργειας. Δεύτερον, οι κανόνες που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική προστασία και οι περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες. Τρίτον, οι διεθνείς περιορισμοί στο εμπόριο και τα προβλήματα που μας τίθενται από τις αμπτυσσόμενες χώρες. Αυτές είναι οι κυριότερες ε, προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Να αναλύσω λοιπόν ένα-ένα αυτά τα τέσσερα σημεία. Τιμές της ενέργειας. Οι διεθνείς ανταγωνιστικές ε, τιμές της ενέργειας και η ε, ασφάλεια της προμήθειας στην ενέργεια είναι πολύ σημαντική για τη χαλιβουργία. δυστυχώ η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου δεν έχουν οδηγήσει σε μείωση των τιμών ενέργειας. Δεν έχουν ανοίξει αρκετά αυτές οι αγορές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κόστος τη ενέργειας είναι περίπου 40% του συνολικού λειτουργικού κόστους των χαλιβουργίων. Ο ηλεκτρισμός και ο οπτάνθρακα είναι οι πιο σημαντικέ πηγέ ενέργεια για την χαλιβουργία, το ΚΟΚ. Οπότε έχει μεγάλο ρόλο το κόστος τους για την παραγωγή των χαλιβουργικών προϊόντων. Πιστεύω και θα θυμάστε κι εσείς ότι ο κύριος Μπούζεκ συνόψισε πάρα πολύ τι πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό στην πρόσφατη έκθεση του. Δεν θα μπω τώρα σε αυτό, σε λεπτομέρειες, αργότερα. Όσον αφορά το δεύτερο σημείο, δηλαδή ε, θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, η περιβαλλοντική μα προστασία είναι απαραίτητη για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και για να λειτουργεί σωστά η νέα αγορά. είναι πολύ σημαντικέ οι περιβαλλοντικέ προδιαγραφέ. Είναι σαφέ αυτό. Η χαλιβουργία παίζει σημαντικό ηγετικό ρόλο, ούτω ώστε να διατηρηθεί η βιωσιμότητα τη ανάπτυξή μα. Διότι εάν χρησιμοποιήσουμε ε, σωστά ε, το χάλιβα, θα έχουμε τρομερές εξοικονομίες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Δηλαδή θα μειώσουμε πάρα πολύ τις εκπομπές. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχει τρομερά καθήκοντα χαλιβουργία και πολλή γραφειοκρατία. Πρέπει να αλλάξουμε τους στόχους της Ένωσης. Αλλά η προσπάθεια να αλλάξουμε συνεχώ του στόχου για να αυξήσουμε την παραβαλλοντική προστασία σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον τομέα. Τι πρέπει να κάνουμε. Την περίοδο μετά 2020 η κλιματική μα πολιτική πρέπει να είναι τόσο ε, διατυπωμένη έτσι ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη συνολικά η κατάσταση της οικονομίας. Και επίσης τα νέα μητρώα για τις διαρροές άνθρακα πρέπει να συνταχθούν με το σωστό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά ορισμένων κλάδων βιομηχανίας και την επίπτωση των τιμών του ηλεκτρισμού. Το τρίτο θέμα είναι οι περιορισμοί στο εμπόριο. Η ευρωπαϊκή χαλιβουργία εξαρτάται προφανώς σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές εμπόριο και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την απελευθέρωση. Η δική μα αγορά χαλιβουργικών προϊόντων είναι από τι πιο ανοιχτέ στον κόσμο, ενώ διάφορε άλλε χώρε εφαρμόζουν διάφορε τρευλώσει και περιορισμού και δίνουν έτσι τεχνητά πλεονεκτήματα στη δική του χαλιβουργία οικονομική κρίση. Εξάλλου, έχει ε, οξύνει ακόμη περισσότερο τα θέματα αυτά. Υπάρχουν μια σειρά από παρεμβάσει από πολλέ χώρε, για παράδειγμα περιορισμοί εισαγωγών, ε, ε, δασμοί, επιστροφές ΦΠΑ, αλλά και άμεσες επιδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ε, δράσει αποφασιστικά κατά του ντάμπινγκ και κατά προϊόντων που έχουν λάβει επιδοτήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε συνεπείς στην αντιμετώπιση μας. Και το τέταρτο φυσικά είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και η χρηματοδότηση της καινοτομίας. Το κύριο πλεονέκτημα της δικής μας χαλιβουργίας είναι ότι έχουμε βελτιωμένη και προωθημένη δομή προϊόντων. Εφόσον όμως ε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τη μείωση των εκπομπών, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε φτάσει στο όριο του τεχνολογικά εφικτού. Δεν θα υπάρξουν ε, νέες τεχνολογίες. Μάλλον αν δεν υπάρξουν νέες τεχνολογικές ε, σοβαρές καινοτομίες και ρήξεις, δεν θα μειώσουμε κατά πολύ περαιτέρω τις εκπομπές. Επειδή οι τεχνολογικές αυτές ρήξεις είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερης έντασης κεφαλαίου, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό και να το ενσωματώσουμε, να το εντάξουμε στο πρόγραμμα 2020. Ε, ε, Αυτοί είναι οι τέσσερις τομείς όπου υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις για τη χαλιβουργία. Είναι σοβαρές προκλήσεις, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να τις αντιμετωπίσουμε, διότι αν δεν τις αντιμετωπίσουμε θα χάσουμε την, ε, το ρόλο μας στην παγκόσμια καλλιβουργία. Η έκθεση πρωτοβουλίας της ΣΥΤΡΕ είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας, να βελτιώσουμε την συμμετοχή μας σε αυτό τον τόσο βασικό, βασικό βιομηχανικό τομέα. Με χαρά βεβαίω θα λάβω υπόψη τις ιδέες και προτάσεις σας και θα προσπαθήσω να τις εντάξω στην έκθεσή μου και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Έχουμε περίπου μισή ώρα στη διάθεσή μας για τη συζήτηση. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούν όλοι να πάρουν το λόγο όσοι θέλουν και η Επιτροπή και να απαντήσει ε, και ο εισηγητής, ο Αντρές Βαρέρα, από το σχέδιο εισηγητής από τους σοσιαλιστές ή κυρία Βαρέρα μάλλον. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Κομισιόν υπέβαλε αυτό το σχέδιο και την στρατηγική για να αναζωογονήσουμε την χαλιβουργία. Ο Χάλιβας είναι στρατηγικός τομέας από οικονομική πλευρά, πολύ σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ο δεύτερος παγκόσμιος παραγωγός 11% ε, όπως είπαμε της παγκόσμιας παραγωγής και έχουμε 360.000 εργαζόμενους. Ο, ο Χάλιβας συγγνώμη, σχετίζεται με πολύ σημαντικές άλλες ε, ε, Πλευρέ τη παραγωγής όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά αλλά όπως είπαμε έχει μειωθεί η ζήτηση κατά 27% και απότομα. Και είναι υψηλή και η τιμή της ενέργειας. Δεν έχουμε λύσει το θέμα αυτό. Και ο ίδιος ο τομέας τη χαλιβουργία πρέπει να κάνει οικονομικές προσαρμογές για να ε, ε, είναι οικολογική και βιώσιμη η δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Η έκθεσή μας λοιπόν είναι σημαντική διότι σημαίνει ότι μπορούμε να θέσουμε ένα όριο προδιαγραφών και χρειάζεται να προσπαθήσουμε να προβλέψουμε την ζήτηση για να προσαρμόσουμε και την προσφορά. Να ξέρουμε δηλαδή τι δημόσια έργα θα έχουμε στο μέλλον στην Ευρώπη όχι μόνο στον τομέα των ε, επικοινωνιών αλλά και των υπηρεσιών όπως είναι τα σχολεία και οι διοικητικές υποδομές να, βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε την εξωτερική αγορά να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός που μας θίγει αλλά να επιμείνουμε οπωσδήποτε εντός της Ένωσης να μην υπάρχουν ε, αθέμητες πρακτικές που αποσταθεροποιούν την αγορά όπως έγινε με την Αρσελό και την Τίσεν. Πρέπει να μιλήσουμε επίσης για όλη την αλυσίδα της παραγωγής, για το κόστος της ενέργειας, που είναι ένα από τα σημαντικά θέματα, να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Να υπάρξουν κριτήρια για την παραγωγή, βράχη και μακροπρόθεσμα, να δούμε και πώς θα υπάρξει καινοτομία, πώς θα έχουμε νέα προϊόντα, βελτιωμένα προϊόντα να προσφέρουμε στην αγορά και την οικονομική πλευρά. Τι θα γίνει με τον ορίζοντα 2020 για τη συνεργασία, για την έρευνα και για τους πόρους της Τράπεζας Επενδύσεων, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις περιοχές που παράγουν χάλιβα. Δηλαδή η έκθεσή μας να μην μείνει χωρίς συνέχεια. Η χαλιβουργία και στην Ευρώπη πρέπει να είναι ανταγωνιστική, βιώσιμη και προσαρμοσμένη. Με μέτρα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Γιατί και βραχυπρόθεσμα, εφόσον έχουμε μείωση 27%, είναι πολύ σημαντική ύφεση από το 2008. Άρα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς, ως σοσιαλιστές, το θέμα των εργαζομένων, το κοινωνικό να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις οι ίδιες στη νέα κατάσταση και επίσης να δουν αν μπορούν να τους βρουν στους εργαζόμενούς τους και θέσεις εργασίας νέες. Συγχαίρω τον εισηγητή, θα υποβάλουμε τροπολογίες για να τη βελτιώσουμε και χαίρομαι που υποβάλουμε αυτή την έκθεση για να μην ξεχάσουμε μια τόσο σημαντική βιομηχανία και να προσπαθήσουμε να, να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο επόμενος συνάδελφος. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραίο είναι που έχουμε μια νέα ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την βιομηχανική πολιτική ε, και την χαλιβουργία που βεβαίως αποτελεί ε, έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ε, πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα είναι ατελείς ε, οι απαντήσεις που έχουμε δώσει στο πρόβλημα αυτό. Ε, η ανακύκλωση και η οικολογική αντιμετώπιση και αυτού του θέματος είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Αλλά και αυτό είναι ε, μερική απάντηση στο πρόβλημα. Το νομοθετικό ε, ε, πλαίσιο δεν είναι φιλικό προς τη βιομηχανία και πρέπει να πούμε ότι ειδικά για το τομέα της χαλιβουργίας είναι ιδιαίτερα εχθρικό και επομένως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τουλάχιστον δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει τούτη τη στιγμή ε, η χαλιβουργία, το κεντρικότερο των οποίων είναι ε, το κόστος της ε, ενέργειας οι Βρυξέλλες παίρνουν αποφάσεις οι οποίες ας πούμε αφορούν περιβαλλοντικές πολιτικές και οι οποίες δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τον τομέα. Ε, και υπάρχει και η πολιτική για την κλιματική αλλαγή που δεν είναι μονάχα ακριβή αλλά είναι και ε, ασταθής. Ε, μην λησμονούμε ότι η Χαλιβουργία αντιμετωπίζει στην Χαλιβουργία η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης είναι μακρά και επομένως θα πρέπει να ληφθούν άλλου είδους λύσεις. Εμείς έχουμε μιλάμε για το σύστημα μετά το αλλάζουμε. Ε, ε, ε, ε, το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, το οποίο το αποφασίζουμε, μετά το αλλάζουμε, το ξαναλάζουμε, όλα αυτά δεν είναι καθόλου θετικά για τον κλάδο. Έναν κλάδο ο οποίος δεν μπορεί πλέον να αναπτυχθεί, γιατί τα μηνύματα των Βρυξελών ε, μπορεί να είναι διαφορετικά από τη μία μέρα στην άλλη ε, και να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στις μονάδες ε, που λειτουργούν. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την, το πρόβλημα του, της ανθρακο, του άνθρακα. Έχουμε ε, το πρόβλημα, την συζήτηση αυτή για τη δέσμευση του, άνθρακα. Ε, όλα αυτά συζητιούνται στις Βρυξέλλες ε, και ξεχνάμε ότι τελικά υπάρχει μεγάλη έλλειψη χρημάτων. Η χρηματοδότηση των ιδεών λοιπόν και των λύσεων δεν μπορεί να γίνει οι κρατικές ε, επιδοτήσεις οι οποίες ε, υπάρχουν σε μερικές ε, χώρες οδηγούν βεβαίως σε στρεβλώσεις της αγοράς αλλά να μην ξεχνάμε ότι η χαλιβουργία δεν αφορά μονάχα μία ή δύο χώρες μέλη. Ε, πρόκειται, για μία, ε, πρόκειται για μία βιομηχανία η οποία αφορά 23 χώρες μέλη. Διαβάζω εδώ διάφορα στην ανακοίνωση της Επιτροπής, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά μπορούν να λύσουν το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πραγματικά ε, το πρόβλημα των, ε, ε, του κόστους της ενέργειας οι χώρες, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε καθόλου να βοηθήσουμε τη Χαλιβουργία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σλάσβος Γκίρεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη κρίση που σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε μία σειρά από μεγάλες προκλήσεις για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το κύριο πρόβλημα. Πριν από ε, λίγο καιρό λέγαμε ότι οι υπηρεσίες ε, θα αποτελέσουν ε, το, το κλειδί για την επιτυχία. Τώρα έχουμε ένα άλλο θέσφατο που είναι οι κλιματικές αλλαγές. Αλλά εντωμεταξύ η χαλιβουργία, η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα πρόβλημα. Έχουμε χάσει το συγκριτικό μας, ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα ε, και αυτό είναι πάρα πολύ κακό για την αυτοκινητοβιομηχανία και για την χαλιβουργία που είναι σημαντικής ε, ε, σημασίας. Ε, βεβαίως ε, είναι γεγονό ότι με τη χαλιβουργία συνδυάζεται και η, η υψηλός βαθμός εκπομπής διοξιδίου του άνθρακο. Απ' την άλλη πλευρά ε, λέμε ότι θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της ε, ανακύκλωσης αλλά νομίζω ότι και όσον αφορά την ε, ανακύκλωση ε, πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις και στο ανακυκλωμένο ε, παλαιοσίδηρο υπάρχει στο σκράπ υπάρχει μεγάλη περιεκτικότητα σε χαλκό και Επομένως ε, ε, δημιουργείται πρόβλημα ε, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το ανακυκλωμένο σίδηρο με μεγάλη περιεκτήρια χαλκού χρησιμοποιείται περισσότερο στην, στον οικοδομικό τομέα. Επομένως υπάρχουν, μην λησμονούμε ότι υπάρχουν και άλλες πρακτικές. Είναι η ΚΒΤΑΦ. Δεν πρέπει να τα λησμονούμε αυτά. Ε, επίσης, να μην ξεχνάμε ότι οι τρίτες χώρες καραδοκούν και περιμένουν ε, να εκμεταλλευτούν αυτήν την ε, ανίσχυρη θέση της Ευρώπης. Μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία και επομένως όλα αυτά που λέγονται από εδώ και από εκεί για κλιματικές αλλαγές και ενέργεια κτλ. δεν θα λύσουν το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μητσιάρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμφωνώ ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του χαλιβουργικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αληθεύει ότι έχουμε καθυστερήσει και περιμέναμε τελευταία στιγμή για να αντιδράσουμε. Τα τελευταία χρόνια είδαμε μείωση 27% στην παραγωγή του τομέα αυτού και ε, ε, απώλεια μεγάλου μέρους του ΑΕΠ μας. Θα θέλαμε λοιπόν να επιδιώξουμε την αύξηση του μεριδίου στο ΑΕΠ του χαλιβουργικού τομέα, ανέκαθεν ναι, αυτός ο τομέας είχε ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Στο μέλλον ούτως ή άλλως θα συζητήσουμε διεξοδικά αυτό το θέμα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα νούμερα που μας έδωσαν οι συνάδελφοι. 177.000 τόνους παράγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δούμε τώρα από ποιοτική πλευρά, προηγούμαστε πάρα πολύ σε σχέση με την Κίνα, παραδείγματος χάρη, και τη δική της παραγωγή. Ο κύριος Γκιούρκ, ε, εξαιρετικός συνάδελφος, μας έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση όλων των προβλημάτων τα οποία καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε και συνόψε την κατάσταση επικεντρώνοντας την προσοχή του σε τέσσερα βασικά σημεία. Ελπίζω να έχουμε την υποστήριξη όλων. Είδαμε τους εμπερικούς περιορισμούς, ε, την τιμή της ενέργειας, τα ε, ρηξικέλευτα τεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται πλέον στον τομέα. Πάνω από 500 μονάδες παραγωγής έχουμε σε 23 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν πρέπει να έχουμε υπερβάλλουσα ε, παραγωγική ικανότητα. Αυτό θα ήταν μια επικίνδυνη τάση. Δεν μπορούμε να επιδιώκουμε την παραγωγικότητα πάση θυσία. Θα πρέπει να επιδιώξουμε αξιοποίηση των πρώτων υλών ε, διότι ο χάλιβας ε, είναι ένα, μια πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας ε, και θα έπρεπε να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Η Ευρωεπιτροπή προτείνει σύσταση μιας ομάδας εργασίας υψηλού επίπεδου η ανταλλαγή των πληροφοριών θα είναι η βάση στην οποία θα εδράζεται το σύστημα, όμως δεν επαρκούν αυτά κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορούμε να σώσουμε την χαλιβουργία χωρίς να κάνουμε και τις αντίστοιχες οικονομικές θυσίε, ε, τις ε, απαιτούμενες επενδύσεις. Για αυτά τα τέσσερα σημεία που εξέθεσε ο κύριος ε, Γκιούρκο, θα έλεγα ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σύστημα στήριξης αρρωγής ε, της ε, Χαλιβουργίας, ο κύριος Σιμάνς και επίσης έκανε ένα εύστοχο σχόλιο διότι μας μίλησε για τις κρατικές επιδοτήσεις που ενδεχομένως συνιστούν στρέβλωση στην αγορά. Όμως ε, Ίσως θα χρειαστεί να κάνουμε μια εξαίρεση για τη χαλιβουργία και να υποστηρίξουμε τον τομέα. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Σλοβακίας. Από το 2012 και μετά βλέπουμε ότι στην χαλιβουργία απασχολούνται πάρα πολλοί άνθρωποι στι μεγάλες μονάδες παραγωγής ε, που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες. Ε, τώρα όμω θέλουν να πουλήσουν ε, τις μονάδες, θα χαθούν θέσει απασχόληση το 2013. Η Σλοβακική κυβέρνηση έδωσε κάποια κίνητρα, έκανε κάποιες παραχωρήσεις και δεν προέκυψαν ως εκ τούτου μαζικές απολύσεις. 260 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημίωση κατεβλήθησαν ε, λόγω της αλλαγής στην κερδοφορία. Ε, τώρα όταν ε, κοιτάζουμε την κατάσταση γενικότερα στην Ευρώπη για να σώσουμε την ευρωπαϊκή χαλιβουργία πρέπει τάχιστα να αναλάβουμε δράση και όπως είπαμε και προηγουμένως ε, στη, στο κατασκευαστικό τομέα και στην αυτοκινητοβιομηχανία η χαλιβουργία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να επιδιώξουμε τις ε, μικρότερες δυνατές εισαγωγές σε χάλιβα από την Κίνα και από την Ρωσία γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να επιδιώξουμε μείωση της παραγωγικής ικανότητας Ίσως θα έπρεπε να επέμβουμε στο, ε, στην πλευρά της ζήτησης. Θα έπρεπε λοιπόν να συμβάλλουμε καταθέτως τροπολογίες για να βελτιώσουμε και το αρχικό κείμενο. Σε κάθε περίπτωση θα προσφέρω την υποστήριξή μου ε, προς τον εισηγητή. Ευχαριστούμε και εσάς. Το λόγο, ε, ε, το λόγο έχει ο συνάδελφος Ρόλε. Κύριοι συνάδελφοι, τρεις σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτον, συγχαίρω τον συνάδελφο Γιούρκ για τη θαυμάσια εργασία που μας υπέβαλε. Δεύτερον, η χαλιβουργία είναι βιομηχανία κλειδί και εδώ θα αποφασίσουμε εάν η πολιτική μας στην Ευρώπη είναι υπέρ ή κατά της βιομηχανίας. Δεν υπάρχει ίσως κτλ. Θέλουμε στην Ευρώπη, στο μέλλον, να έχουμε βιομηχανίες και όχι διακηρύξεις υπέρ της βιομηχανίας. Τότε πρέπει να λάβουμε και τα αναγκαία μέτρα που θα έχουν τι αναγκαίες επιπτώσεις. Διότι η χαλιβουργία δεν είναι μόνο οι διάφορες μονάδες χαλιβουργίας. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο. Και τρίτον, γι' αυτό το θέμα φαίνεται ποιες, ε, πόσο τρομερές θα μπορούσαν να ήταν οι αποφάσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής. Εάν οι επιβαρύνσεις της στη βιομηχανία είναι τόσο συνεχείς και αυξάνονται, τότε ε, πολύ δύσκολα θα επιβιώσουν διάφορα βιομηχανικοί κλάδοι και άρα και θέσεις εργασίας τους. Μόνο δύο απαντήσεις είναι δυνατές. Πρώτον, δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνουμε τόσο πολύ τις βιομηχανίες, να μειώσουμε καλύτερα την επιβάρυνση και δεύτερον, οι ειδικέ ρυθμίσεις που έχουμε δημιουργήσει πρέπει να τεθούν ε, υπό συζήτηση και πάλι. Δεν είναι δυνατόν να τους πιέζουμε και από τις δύο μεριές. Διότι αν τους πιέζουμε τόσο πολύ, άμα λέμε τόσα ψέματα, χάνουμε τις θέσεις εργασίας. Πρέπει λοιπόν ως Επιτροπή Βιομηχανίας να πούμε ξεκάθαρα τι θέλουμε. Ήρθε η ώρα πιστεύω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μία προσπάθεια να ενισχύσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία έντονη. Εάν θέλουμε να έχουμε θέσει εργασία για να έχουμε και φορολογικά έσοδα από τι θέσει εργασία, για να έχουμε κοινωνική πολιτική, πρέπει να βοηθήσουμε τη βιομηχανία. Δεν γίνεται χωρί σαφή ενίσχυση τη βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Γκέμπελ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, σε 15 χρόνια το βάρος της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έπεσε από το 20% στο 15%. Και αυτό είναι ένα πραγματικό στοιχείο. Σε πολλούς τομείς βλέπουμε να κλείνουν εργοστάσια, να μειώνουν το προσωπικό, να έχουν απολύσεις και επίσης πολλές είναι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες οι οποίες αποφασίζουν να φύγουν εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία από τις βιομηχανίες αυτές, αλλά είναι στρατηγική σημασία, είναι και η χαλιβουργία. Ο εισηγητής έχει απολύτως δίκιο όταν ε, λέει ότι πάντα θα έχουμε ε, όπως και αν είναι το μέλλον μας, θα χρειαζόμαστε και, και χάλιβα και χιτοσίδηρο και όλα αυτά τα προϊόντα της ε, χαλιβουργίας. Το πρόβλημα όμως στην χαλιβουργία είναι ότι βοηθούντος και του κλίματος και των τεχνολογικών εξελίξεων χρειαζόμαστε λιγότερο χρόνο. Για να ξανακατασκευαστεί ο πύργος του Άιφελ σήμερα θα χρειαζόμαστε πλέον μονάχα το 1 τρίτο του χάλιβα που χρησιμοποιήθηκε στην εποχή της κατασκευής του. 1 τρίτο, 1 τρίτο. Αυτό είναι συνώνυμο της πρόοδου βέβαια στην μεταλλουργία. Τα προβλήματα όμως της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δεν είναι αυτά που λέμε τώρα και πολύ σωστά το ανέφερε ο συνάδελφος Γκύρικ. Ε, το πρόβλημα είναι το μεγάλο κόστος της ενέργειας, ε, τα, το περιβαλλοντικό βάρος, ε, δηλαδή των περιβαλλοντικών κανόνων, που δεν βαραίνει τη χαλιβουργία της Κίνας ή των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθούν να επενδύουν ε, οι χαλιβουργίες, αλλά εκτός Ευρώπης. Η Arcelor Mittal ε, συνεχίζει τη στην Αφρική, στην Νότια Αμερική, στην Ασία, αλλά κλείνει ε, τα εργοστάσια στην Ευρώπη. Και δεν είναι η μόνη. Συνάντησα πρόσφατα τον δόκτωρα Χέντερ, ο οποίος είναι η σκεπτόμενη κεφαλή του τρίτου κατασκευαστή στην Ευρώπη κατασκευάζουν νέο εργοστάσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και θα παράγουν πρώτη ύλη για τις βιομηχανίες στην Ευρώπη. Και είναι πολύ απλό. Γιατί το κόστος στην ενέργεια, ε, το κόστος της ενέργειας είναι πολύ χαμηλότερο εκεί. Το κόστος της ενέργειας είναι μεγαλύτερο στη χαλιβουργία από το κόστος της εργασίας και από το μισθολογικό κόστος και επομένως ε, ε, τι να σας πω τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε ας πούμε ε, άλλου είδους πολιτική δεν θέλουμε να επενδύσουμε στο σχιστολιθικό αέριο γιατί έχουμε διάφορες ιδεολειψίες τις οποίες δεν έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείες και έχουν μειώσει το κόστος της ενέργειας. Ένας παραγωγός ε, ε, σωλήνων ε, στην Γαλλία αποφάσισε και αυτός να μετακινήσει την παραγωγή του στις ΗΠΑ λόγω ακριβώς του κόστους της ενέργειας. Και τώρα θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη. Λες και έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Στην Στοκχόλμη το ΖΙΕΚ ε, είχε μεγάλη δυσκολία να εξηγήσει ότι ε, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως λέμε όσον αφορά τις κλιματικές ε, αλλαγές. Εμείς παρόλα αυτά λέμε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Έχουμε βάλει λάβαρο το Κιώτο και λέμε ότι πρέπει διαρκώς να μειώνονται οι εκπομπές, ενώ το ΖΙΑΚ είπε ότι δεν είναι το κύριο πρόβλημα οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Στην Αυστραλία η ε, κυβέρνηση έκλεισε μια ύπατη που είχε δημιουργήσει ε, για την κλιματική αλλαγή. Την έκλεισε, τελεία και παύλα. Και είμαι σίγουρος ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και η Αυστραλία ακολουθούμενη και τους Νεοζηλανδούς και, ε, θα, και τους υπόλοιπους θα βγουν και από τη Συμφωνία του Κιώτο. 11% ε, ε, ε, των συνολικών εκπομπών των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος ε, παράγονται από τη χαλιβουργία. Εσείς πιστεύετε ότι αν μειώσουμε ε, κατά 20% τις εκπομπές αυτές ε, θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε την Κίνα ή τις Ηνωμένε Πολιτείε. Κοιτάξτε, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε γύρω από τον άνθρακα και το χάλιβα. Και εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των χωρών της θέλει να παραμείνει ηγέτιδα στην, της βιομηχανίας, τότε θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε διαρκώς να πιέζουμε ε, τις, ε, τη βιομηχανία μας και όχι μονάχα τη χαλιβουργία με τέτοια κόστη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Είδα ότι προσθέθηκαν αγορητές στον κατάλογο ε, και εγώ ε, για το λόγο αυτό <clears throat> και για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα μιλήσω εγώ η ίδια. Ε, όμως σε αυτό το τελευταίο τμήμα της συζήτησης θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μην ξεπεράσετε τα δύο λεπτά, να μην μακρηγορήσετε γιατί διαφορετικά θα ξεπεράσουμε τον προβλεπόμενο χρόνο. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον επόμενο συνάδελφο Χένινγκ, Κρόιτσμαν ε, και μετά ο ε, εισηγητής. Χένινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, εγώ θα μιλήσω δύο λεπτά, αλλά μετά δύο λεπτά, την επόμενη φορά να μιλήσουν δύο λεπτά όλοι. Είναι θέμα δικαιοσύνη. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Ρόλ και εν μέρη με αυτά που είπε ο κύριος Γκέμπελς. Ναι, βεβαίως Έκλεισε το μικρόφωνο του κύριου Ενέν. Ε, ναι, βεβαίως χρειαζόμαστε ισχυρή χαλιβουργία στην Ευρώπη γιατί δημιουργεί θέσεις εργασίας και καλές θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενε οι οποίες ε, ε, επανατοποθετούν στον κλάδο τον παραγόμενο πλούτο. Απ' την άλλη πλευρά όμως πρέπει να πούμε ότι και η βιομηχανία γενικότερα και η χαλιβουργία δεν ε, έχει πρόβλημα λόγω του υπερβολικού κόστους. Ε, έχει πρόβλημα λόγω της, ε, του στραβλωμένου ανταγωνισμού από την, τις αναδεόμενες χώρες. Στη Γαλλία, ας πούμε, ήρθε η Αρσελόν Μιτάλ. Πιστεύετε ότι η γαλλική χαλιβουργία δεν μπορεί να παράγει σε ανταγωνιστικές τιμές για να κερδίσει τιμές. Βεβαίως μπορεί, αλλά η στρατηγική του κυρίου Μιτάλ ήταν διαφορετική. Αγοράζει επιπιστώσει η ε, ε, επιπιστώσει. Ε, προσπαθεί να αντλήσει όλο το δυναμικό των εργαζομένων, όλων των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της έρευνας και μετά να τα πάρει και να τα πάει αλλού. Εάν είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό που, αυτό που δημιουργεί πρόβλημα στην γαλλική σιδηρουργία, αν το πιστεύουμε ακόμα δηλαδή ότι είναι το μεγάλο κόστος, τότε κάνουμε μεγάλο λάθος. Ξέρουμε ότι αυτή αυτή τη στιγμή η Μιτάλε θέλει να κλείσει τις υψηκαμίνους στη Γαλλία για να, πάει στην, να τις πάει στην ε, ε, Ινδία. Μιλάμε εδώ όχι μονάχα για την χαλιβουργία και τη σιδηρουργία, μιλάμε όπως έχει υποθεί πολλές φορές εδώ και για ε, άλλες βιομηχανίες, την αεροναυπηγική, την αυτοκίνητο βιομηχανία. Μιλάμε δηλαδή στο σύνολο για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων ε, που ε, ε, θα χάσουν οπωσδήποτε τη δουλειά τους γιατί είναι στοχευμένες οι επιθέσεις κατά της χαλιβουργίας. Και βεβαίως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εμποδίσουμε αφενός τον κύριο Μιτάλ να φύγει και να πάει να εκμεταλλευτεί άλλους εργαζόμενους στον τρίτο κόσμο, αλλά κυρίως να βοηθήσουμε τους δικούς μας εργαζόμενους. Ευχαριστώ κύριο Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο Σάνφος Ρόιλ. Μία σύντομη παρατήρηση. Η γερμανική χαλιβουργία δεν παράγει μόνο χάλιβα, παράγει λύσεις για τους πελάτες της. Αν το βγάλουμε αυτό από την εξίσωση, ορισμένοι λένε είναι εντατική ενέργειας, ε, αν είναι μόνο αυτό το θέμα μπορούμε να εισάγουμε χάλιβα εκτός Γερμανίας, αλλά από ε, το εξωτερικό στη Γερμανία. Αλλά αυτό θα ήταν λάθος. Το θέμα είναι ότι η χαλιβουργία μας παράγει προσαρμοσμένα για τους πελάτες της προϊόντα. Υποστηρίζω όλους που λένε ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρώπη ως βιομηχανία πρέπει να υπάρχει ανταγωνιστική χαλιβουργία. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και λογικές τιμές ενέργειας γιατί αλλιώς δεν μπορούν να συνεχίσουν να επιβιώνουν αυτές οι επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Λάνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε δίκες. Το πλαίσιο δεν πρέπει να επιδεινωθεί για, τον, ε, για τη χαλιβουργία, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι ότι έχει μειωθεί κατά πολύ η ζήτηση. Το 2007 στην Ευρώπη ε, είχαμε 14,7 νέα αυτοκίνητα, νέε άδειε αυτοκινήτων, ενώ φέτο έχουμε 11,2. Αυτό σημαίνει ότι παράγουμε λιγότερα αυτοκίνητα. Ή στον κατασκευαστικό τομέα είναι ακόμη πιο δραματική η κατάσταση. Η ζήτηση για κατασκευαστικό άνθρακα είναι το 30% της ζήτησης πριν από την κρίση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει ζήτηση για χαλιβουργικά προϊόντα. Πρέπει να ενισχυθεί αυτή η ζήτηση. Και δεύτερον, το μεγάλο πρόβλημα των ανταγωνιστών μας. Έχουμε πολύ περισσότερους ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά. Έχουμε νέα χαλιβουργία στο Αμπουντάμπι που εισάγουν στην Ευρώπη, στη Ρωσία και, και στην Τουρκία επίσης. Πολύ ισχυροί ανταγωνιστές. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτούς τους δύο παράγοντες. Πρέπει να ενισχυθεί η ζήτηση για χαλιβουργικά προϊόντα και να ενισχυθεί η καινοτομία ούτω ώστε να επικρατήσουμε έναντι των ανταγωνιστών. Να αυξήσουμε δηλαδή την ανταγωνιστικότητα. Βεβαίω και το θέμα των τιμών τη ενέργεια είναι στο πλαίσιο. Αλλά πολύ αποφασιστικά είναι και τα ζητήματα τη έρευνα και ανάπτυξη γιατί χρειαζόμαστε προϊόντα που να είναι υψηλά υψηλή τεχνολογική αξία τα προϊόντα, ούτω ώστε να είναι καλύτερα από αυτά που εισάγονται από τη Ρωσία. Και αν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή στη δομή, αυτό έχει να κάνει και με τους εργαζόμενους. Θα ήθελα το μοντέλο της ΕΚΑΧ που ήταν τόσο επιτυχές και ανάπτυξε τον άνθρακα και το χάλιβα για 50 χρόνια να το αξιοποιήσουμε, να υπάρχει κοινωνικός διάλογος μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών, της Κομισιόν για να γίνει η αναδιάρθρωση της χαλιβουργίας από κοινού ούτως ώστε να μην μείνει κανείς στο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Σνάλφο Γκέμπελ για αυτά που είπε. Υποστηρίζω όλα αυτά που υπόθηκαν. Και τον Σνάλφο Κρόιτσμαν βεβαίω που υποστήριξε τον Σνάλφο Γκέμπελ και τον Σνάλφο Ρόιλε. Εάν θέλουμε χάλιβα στην Ευρώπη θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα του υψηλού κόστους ενέργειας. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν αλλά δεν είναι μόνο θέμα της χαλιβουργίας και άλλοι τομείς ε, εγκαταλείπουν ε, την Ευρώπη και πηγαίνουν σε άλλες περιοχές. Στη δική μου περιφέρεια βλέπουμε ότι τα νέα αυτοκίνητα παράγονται όλο και περισσότερο αλλού. Πρέπει πραγματικά να ανοίξουμε τα μάτια μας, να μην κρυβόμαστε από την πραγματικότητα. Αυτά τα θέματα δεν θα συμβούν στο εγγύς μέλλον, συμβαίνουν ήδη. Και αυτό που ανάφερε ο συνάδελφος Γκέμπελς. Πρέπει οπωσδήποτε πρέπει να δούμε τη σύνδεση κλιματολογικής αλλαγής και ενέργειας, ούτως ώστε μακροπρόθεσμα να μην ανήκουμε στους χαμένους αλλά στους κερδισμένους. Υπογραμμίζω αυτό που είπε και ο συνάδελφος Κρόιτσμαν. Το θέμα είναι να δημιουργούμε προϊόντα υψηλής αξίας. Αν δεν έχουμε τέτοια προϊόντα, τότε θα μειωθεί και η έρευνα. Αν όχι σήμερα, αύριο, οπότε όλοι οι κλάδοι της βιομηχανίας μέσο και μακροπρόθεσμα θα υποφέρουν. Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει επιγόντως να μας απασχολήσουν. Ευχαριστώ το θαυμάσιο κείμενο του συγητή και θα υποστηρίξω την εργασία του και ευχαριστώ. Να σας πω ότι θα κλείσω τον κατάλογο των αγοριτών γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Ρούμπικ, Περτσίνα, Τρότμαν. Και βεβαίως θα επανέλθουμε στο θέμα όταν θα συζητήσουμε τις τροπολογίες και θα μπορέσετε να ξαναπάρτε το λόγο, Ρίπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Περί τίνος πρόκειται. Εάν θέλουμε να καταναλώνουμε στην Ευρώπη πρέπει να δούμε και τι παράγουμε. Και φυσικά πρέπει να έχουμε μια αλυσίδα που να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας. Α, και εδώ βεβαίως παίζει ρόλο η τιμή των πρώτων υλών, η τιμή της ενέργειας, ε, το εργατικό κόστος που είναι πολύ υψηλό στην Ευρώπη σε σχέση με άλλες περιοχές. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την παραγωγή μας πρέπει να δούμε τη στρατηγική μας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ισχυρό ανταγωνισμό. Τον παγκόσμιο. Για να επερασπίσουμε την παραγωγή μας. Οπότε, άλλοι στην Ευρώπη δημιουργούν ένα τέτοιο κλίμα, όπως πολλές ε, μη κάπα όμικρον, που έχουν θέσει ως στόχο να διώξουν με διάφορες δράσεις τη βιομηχανία από την Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν να τους επιτρέψουμε να κάνουν αυτό το πράγμα. Πρέπει να έχουμε σοβαρή βιομηχανική πολιτική και καλό την Επιτροπή Ήτρε να κάνουμε μια μελέτη, να δούμε ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις που θέλουν να διώξουν την παραγωγή από την Ευρώπη και να επανέλθουμε σε ένα πολύ χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρόλα αυτά που είπαμε για τις νέες τεχνολογίες, για την ανάπτυξη και για τα χαρακτηριστικά του χαλιβουργικού τομέα, εξυπακούεται ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ενεργοβόρος ο τομέας. Όμως, εάν δεν δημιουργηθούν ικανοποιητικές προϋποθέσεις και να έχουμε τις ίδιες τιμές ενέργειας όπως και στον υπόλοιπο κόσμο, τότε είναι πολύ απλό, θα φύγει το κεφάλαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συχνά αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα της δαπάνες λόγω υψηλών τιμών ενέργειας. Αυτό έχει ιδιαίτερα ερνητικέ επιπτώσεις στη βιομηχανία μας. Από τεχνολογική σκοπιά πρέπει να χειριστούμε το θέμα τόσο ώστε οι δικοί μας παραγωγοί να έχουν τις ίδιες τιμές. Όπως τις είπα και στην Κίνα, Αλλιώς ποτέ δεν πρόκειται να διατηρηθεί η χαλιβουργία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Τρουθμάν. Ευχαριστώ, αγαπητή Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συμφωνήσω απολύτω με αυτά που είπε ο συνάδελφος Γκέμπελς, ε, ο οποίο ήταν μάλιστα μεταξύ των βουλευτών που συμμετείχαν στην πλατφόρμα ε, την γαλλο-λουξεμβουργική, βέλγο-γαλλο-λουξική Λουξεμβουργική Πλατφόρμα για την Ασαρόλ Μετά. Επίσης ε, ε, ε, πρέπει να σας πω ότι μπορεί να μην συμφωνώ με τον κύριο Ενέν γενικά, αλλά με την ανάλυση του, γιατί είναι γεγονός ότι θα πρέπει να βρεθούν οι πόροι αυτοί οι οποίοι είναι απαραίτητοι για όλο τον κλάδο, γιατί μιλάμε εδώ για ευρεσιτεχνίες, για διπλώματα ευρεσιτεχνιών, τα οποία αφορούν όλο τον κλάδο της χαλιβουργίας. Πρέπει να έχουμε μια πολύ σημαντική ε, πολιτική, σοβαρή πολιτική, κατανοώντας ε, ότι όλη η παραγωγική ε, οικονομία της Ευρώπης εξαρτάται από, τη, από τον Χάλιβα. Μια βιομηχανική στρατηγική είναι πάρα πολύ σημαντική, πέρα από τη συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε για τη χρηματοδότηση, για τα κεφάλαια κτλ. Ξέρουμε τι συνέβη με τον με το κόστος του άνθρακα. Ξέρουμε τι, έγινε με την, τι γίνεται με την εξέλιξη των τεχνολογιών που αφορούν τον άνθρακα, την αποθήκευσή του κτλ. Δεν πρέπει ε, να ε, μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε ε, να συνδέουμε τα πάντα με την χαλιβουργία και όλο το κόστος τελικά της έρευνας να βαραίνει τη χαλιβουργία. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Ματία Πελεγκρίνη Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριε Πελιγκρίνη, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί ακούσαμε πολλές παρεμβάσεις ούτως ή άλλως. Επιτρέψτε μου να πω πρώτα απ' όλα, ε, να εξηγήσω μάλλον τον λόγο για τον οποίο ε, οδηγηθήκαμε στην ε, κρίση. Νομίζω ότι οι βουλευτές που πήραν το λόγο αναφέρθηκαν σε διάφορους λόγους, λέγοντας αυτός είναι ο κύριος λόγος, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για μία σειρά λόγων που οδήγησαν στην κρίση σε συνδυασμό βέβαια και με την χαμηλή ε, ζήτηση ε, και αυτό αναφέρθηκε από τους βουλευτές και είναι σίγουρα ένα μεγάλο ε, πρόβλημα. Κάτι άλλο το οποίο αναφέρθηκε εδώ είναι η στρέβλωση του ανταγωνισμού και αυτό το έχουμε καταγράψει <clears throat> στην ανακοίνωσή μας. Βλέπουμε επίσης όλο και πιο πολλές περιοριστικές εμπορικές ε, ε, πρακτικές ε, οι οποίες δυσχεραίνουν την κατάσταση. Άλλοι μεταξύ μόνοι είπαν ότι η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή βάρινε πολύ. Βλέποντας όμως το σχέδιο δράσης θα διαπιστώσετε ότι η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι προτίθεται να κάνει ένα κοινό σχέδιο δράσης κτλ. Αυτό έχει γίνει πλέον, είναι πραγματικότητα. Ε, και ε, στην ε, DG Enterprise, στον ιστότοπο που έχει DG Enterprise μπορείτε να δείτε ε, θα δείτε επίσης ότι το κόστος ε, της ε, ρύθμισης για το ξεπέρασμα των κρίσεων τύπου της κρίσης του 2009 βάρινε πολύ στην βιομηχανία. Πρέπει να πω λοιπόν ότι όλα αυτά που είπατε είναι σωστά, απλώς το πρόβλημα προέκυψε από ένα συνδυασμό όλων αυτών που αναφέρατε. Να πω τώρα δύο λόγια σχετικά με την εργασία του εισηγητού. Ο εισηγητής λοιπόν ε, ε, έκανε, ανέφερε τέσσερα κεφάλαια στην εργασία του, τα οποία ε, είναι σωστά. Εγώ θα έλεγα όμως ότι υπάρχει και ένα πέμπτο κεφάλαιο, που είναι η κοινωνική διάσταση, όπως θα έχετε δει και ε, πολλοί βουλευτές αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό, δηλαδή ε, σε, σε κλεισίματα εργοστασίων ε, που έγιναν ή πρόκειται να γίνουν σε διάφορες χώρες μέλη. Αλλά βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί αυτή η αναδιάρθρωση που λαμβάνει η χώρα στην Χαλιβουργία. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ε, ε, να χρησιμοποιηθούν ε, τα χρήματα για κατάρτιση και επανακατάρτιση. Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι, μεγάλη, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης δεξιοτήτων ε, στον τομέα. Τέλος, να πω δύο πράγματα ακόμα. Ένα σχόλιο για την κλιματική αλλαγή. Ε, όλοι ε, εξηγήσατε το κόστος το οποίο αφορά την κλιματική αλλαγή και βαραίνει την ε, χαλιβουργία. Υπάρχει ένα θετικό με το ΣΕΔΕ στην ανακοίνωση της Επιτροπής θα δείτε ότι καλούνται τα κράτη-μέλη ε, να ε, ε, ταυτοποιήσουν την πραγματική χρήση του, ΣΕΔΕ. Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα να, πείτε, να πούν τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν τα χρήματα τα οποία έχουν προκύψει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτό είναι ένα κίνητρο το οποίο σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει μάλιστα και υποχρεωτικό, γιατί αυτά τα χρήματα ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έρευνα στην βιομηχανία. Ε, τελευταία μου ε, σκέψη. Ε, όσον αφορά την βιομηχανία, την ενέργεια βιομηχανία. Εμεί, ε, σαν ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον ορίζοντα 2020 έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουμε κάποιε εταιρικέ σχέσει οι οποίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ η Spiring Miri, ε, η οποία είναι, ε, ε, είναι διαδικασίες που μπορούν να προωθήσουν την εταιρική σχέση μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου. Αυτά και ευχαριστούμε και τον εισηγητή για το όσο ανέφερε στην έκθεσή του. Ευχαριστούμε, Δ. Πελεγκρίνη. Πολλά μα είπατε και ενδιαφέροντα, παρά το λίγο χρόνο που είχατε στη διάθεσή σα, λέει η πρόεδρο. Θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή τώρα, έτσι ώστε να κάνει κάποια τελικά συμπεράσματα, ε, σας βεβαίω ότι θα επανέλθουμε στο θέμα και θα έχει τη δυνατότητα να ξαναμιλήσει. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Με μεγάλη μου χαρά θα απαντούσα σε κάθε ερώτημα ξεχωριστά, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό σήμερα. Δώστε μόνο την ευκαιρία να απαντήσω στον κύριο Ρόιλ. Μας είπε ότι μπορούμε να έχουμε μία ε, προσέγγιση ε, με ενδιασμούς ε, για τη χαλιβουργία. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για τους σκοπούς μας. Βλέπουμε το περιεχόμενο της έκθεσης και το μέγεθος των προκλήσεων και αυτό ξεκάθαρα καταδεικνύει ότι η Επιτροπή Ήτρε θα σταθεί στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Χαλιβουργίας και με τις παρεμβάσεις που άκουσα κατάλαβα ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, στις υψηλές τιμές ενέργειας, στη γραφειοκρατία, στους εμπορικούς περιορισμούς, στη χρηματοδότηση πρωτοβουλειών έρευνας και τεχνολογίας. Επίσης θα συνεκτιμήσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις κάθε παράγοντα ξεχωριστά, όπως μου ζήτησαν τα μέλη της Επιτροπής. διότι αυτός ο βιομηχανικός ε, κλάδος ε, είναι η βάση της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει αυτόν τον τόσο σημαντικό ρόλο και περιμένω με ανυπομονησία τις εισηγήσεις των συναδέλφων και θα τις συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών η 13η Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Ήτρα θα λάβει χώρα την 16η Δεκεμβρίου. Ευχαριστούμε. Θα περάσουμε στο δεύτερο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Όπως σας είπα στην αρχή έχει γίνει μια αντιστροφή στο πρόγραμμα, έγινε μια αλλαγή στη ημερησία διάταξη Τη πρωινή συνεδρία, επομένω θα δώσω αμέσως το λόγο στον δόκτωρα Βιόλα για να μας ε, παρουσιάσει αυτήν την δέσμη η οποία έχει δημιουργήσει μεγάλη ανυπομονησία και προσδοκίες στα κράτη-μέλη. Ε, θα έχετε όλο το χρόνο στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές. Είναι μεγάλη μου τιμή που ήρθα σήμερα για να σας παρουσιάσω για πρώτη φορά τον ε, κανονισμό για την συνδεδεμένη Ήπειρο και το πακέτο μέτρων ε, που υιοθετήθηκε μαζί με την ανακοίνωση, δηλαδή σύσταση της 11 η Σεπτεμβρίου για αυτό το ζήτημα. Είναι μεγάλη μου χαρά πραγματικά, διότι μου δίνεται η ευκαιρία να σας εξηγήσω βήμα προς βήμα ε, τη διάρθρωση του κανονισμού. Είναι η πρώτη μας ε, επαφή, το ανέφερα, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία, είμαστε στη διάθεσή σας για να παράσχουμε η αδίποτε πληροφορία ή διευκρίνηση επιθυμείτε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε το ιστορικό υπόβαθρο. Για ποιο λόγο ποιο είναι ο λόγο ύπαρξη του κανονισμού και αν κοιτάξουμε την ε, ευρύτερη εικόνα τη ανάπτυξη ε, των νέων ε, τεχνολογιών πληροφορία και τη συμβολή του στου βιομηχανικού τομεί ευρωπαϊκή οικονομία. Έχουμε κάνει μία διεξοδική ανάλυση του ψηφιακού θεματολογίου επικεντρωνόμενη στους βασικούς μας στόχους 360 μοίρες αλλαγή πορεία, ή μάλλον ε, εξετάζουμε σφαιρικά το ζήτημα, ούτω ώστε να καλύψουμε όλους τους τομείς που επηρεάζονται από τις νέες τεχνολογίες. Η βασική υποδομή και κυρίως ο κανονισμός για τις υποδομές είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι στα πλαίσια του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου καταλήξαμε συμφωνία και η προτινόμενη χρηματοδότηση μειώθηκε σε ένα κονδύλι ενός δις για τη νέα έρευνα ε, οπότε για την ε, επερχόμενη περίοδο, εκτός και αν υπάρξει αναθεώρηση, δεν θα προσφερθεί δημόσια χρηματοδότηση για, την, για τα δίκτυα αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να εισρέψουν ιδιωτικά ε, κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της έρευνας ε, και καταλαβαίνετε ότι έως εκ τούτου αποκτά και μεγάλο βάρος ο κανονισμός. Ε, σε σχέση πάλι με, την, με το ψηφιακό θεματολόγιο μιλάμε για την αναμόρφωση των δημοσιών υπηρεσιών. Τι μπορεί να προσφέρουν νέες τεχνολογίες στις δημόσιες υπηρεσίες για να είναι πιο αποτελεσματικές, πιο ποιοτικές για τους πολίτες ε, και αντί να επισύρουν απώλειες, ε, να επιφέρουν κέρδη. Ε, μιλάω για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μπορεί να μας προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος και μπορεί να προσφέρει στους πολίτες πιο συγκεκριμένα. Τώρα, δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης. Ένα εκατομμύριο θέσεις έχουμε στον τομέα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και αν λάβει κανείς υπόψη ότι έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με την ανεργία των νέων, είναι παράδοξο να το παρατηρούμε ταυτόχρονα με τις σωστές ψηφιακές δεξιότητες υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για τους νέους. Έχουμε την ανακοίνωση για την ανοιχτή εκπαίδευση, την παρουσίαση σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται για την τροποποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην Ένωση. Οι δεξιότητες είναι λοιπόν στον πυρήνα ε, του συνολικού ε, οικοδομήματος μιας ε, πιο αποτελεσματικής και σύγχρονης εξυγχρονισμένης τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε ασφαλή δίκτυα, χρειαζόμαστε κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα, κυρίως για το μέλλον, το υπολογιστικό νέφος που είναι απαραίτητο για την παροχή των διακυβευόμενων υπηρεσιών. Το Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει συγκεκριμένα μέτρα και σε τρει εβδομάδες τον Οκτώβρη για πρώτη φορά θα εξετάσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την ψηφιακή ενιαία αγορά, την πρόοδο σε σχέση με την ε, ενιαία αγορά των τηλεπικοινωνιών επίσης. Ε, προ... κατά την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, προετοιμάσαμε συγκεκριμένα μέτρα, αυτό μας είχε ζητηθεί, ούτω ώστε να υλοποιήσουμε το βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για να επιτύχουμε τους στόχους μας σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, διότι όπως σας είπα και στην αρχή είναι κέρια σημασία σε αυτό για την τόνωση της ανάπτυξης, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ε, της Ευρώπης, κυρίως σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Το πακέτο που εγκρίθηκε στις 11, όπως σας είπα στην αρχή, συναπαρτίζεται από τρία τμήματα. Έχουμε μία ανακοίνωση που θέτει το όραμα για την ενιαία ψηφιακή αγορά τηλεπικοινωνιών ε, και ορίζει ένα σειρό βημάτων ε, που πρέπει να πραγματοποιηθούν με τρόπο ώστε να υπάρξει πλήρης ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Επίσης, καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης, μία οδηγία με τις βέλτιστες πρακτικές, δηλαδή με τρόπο ώστε να έχουμε σταθερότητα και νομική ασφάλεια για τον κανονισμό, για την πρόσβαση κυρίως στα ευρυζωνικά δίκτυα και ο προτινόμενος κανονισμός για τη συνδεδεμένη ήπειρο που θα είναι και το αντικείμενο της σημερινής μου παρουσίασης. Τι προτείνουμε, ας κοιτάξουμε πρώτα απ' όλα τον κανονισμό. Σας είπα και στην αρχή ότι είναι το γερό θεμέλιο των υποδομών. Χωρίς τις υποδομές δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Αυτό είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους ...αν δεν έχουμε ευρυζωνικές υποδομές. Δεν μπορούμε να έχουμε ψηφιακές τάξεις αν δεν έχουμε ευρυζωνικές υποδομές. Δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά δεδομένα πάλι αν δεν υπάρχει διασυνδεσιμότητα. Η διασυνδεσιμότητα είναι η κόλλα που ε, τα ενώνει όλα δεν ε, μπορούμε να προσφέρουμε προηγμένες υπηρεσίες αν δεν υπάρχει αυτό. Είναι προϋπόθεση βασική και στην Ευρώπη ποικίλη κατάσταση σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε κάποιες χώρες που είναι στην κορυφή του κόσμου για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και άλλοι, άλλες χώρες που είναι ουραγοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η διάσταση που μας έχει ξεφύγει διότι αν κοιτάξουμε τη δική μας διασυνδεδεμένη ήπειρο των 500 εκατομμυρίων πολιτών καταλαβαίνουμε ότι είναι η ενδυνάμει πρώτη παγκόσμια ε, διασυνδεδεμένη αγορά κοιτάξετε παραδείγματο χάρη του λίγου ευτυχισμένου που υπάρχουν ε, δεν ε, αποτελούν μια κρίσιμη μάζα για να μπορέσουμε χρησιμοποιώντα του να ανταγωνιστούμε στην παγκόσμια σκηνή και δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη διαδικασία που θα δημιουργήσει νέε θέσει απασχόληση. Γι' αυτό θέλουμε κλίμακα, η ε, οικονομία κλίμακα σε, ολόκληρη την γυραιά Ήπειρο ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια έγκυρη πρόταση και να φτάσουμε στην πρώτη γραμμή και να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο. Ε, φυσικά αυτό θα πρέπει να είναι επωφελές για τους πολίτες. Ε, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να εξετάσουμε μόνο την, ε, το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αλλά να κοιτάξουμε και θα προσφέρει διασυνδεμένη ήπειρο στους πολίτες. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να προσφέρουμε ανοιχτές υπηρεσίες, ανοιχτό διαδίκτυο, διαδικτυακή πρόσβαση μάλλον, ανοιχτά δίκτυα, εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Η πρόταση που κάνουμε είναι ιδιαίτερα ισοσκελισμένη. Βασικά εδράζεται ε, επί τριών πυλώνων και ε, υπάρχει μια, ε, ένα νήμα της Αριάδνης που διατρέχει το σύνολο των ιδεών. Δεν έχουμε κάνει μια τυχαία συλλογή ιδεών μέσα σε ένα προτινόμενο νομοθέτημα. Υπάρχει ιδιαίτερη συνοχή. δούμε το πρώτο σκέλος. Ε, ή μάλλον αν αφαιρέσουμε οποιοδήποτε σκέλος τότε καταρρεί ολόκληρη η πρόταση. Ε, ποια είναι η λογική που κρατάει τη συνοχή του πακέτου ε, χρειαζόμαστε μια ασφάλεια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε σχέση με το ποιος είναι ο εφαρμοστέος κανονισμός, ποιο είναι το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο και τι έχουν να κερδίσουν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την συνεισφορά της βιομηχανίας ε, για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών το πλέον σημαντικό για να έχουμε το διασυνδεδεμένο φάσμα είναι ότι όταν είναι διαθέσιμο το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων θα πρέπει να ξέρουμε ε, σε ποια τιμή θα είναι διαθέσιμο και πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμο. Χρειαζόμαστε ασφάλεια σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των ε, δικτύων ε, επίγειων ή ασυρμάτων και μείωση φυσικά της γραφειοκρατίας που συνοδεύει όλα αυτά τα μέτρα. Ένα άλλο στοιχείο που επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι η πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα και αν επιθυμείτε ε, πρόσβαση σε υπηρετική κλίμακα θα πρέπει εικονικά να διασυνδεθούν όλα αυτά τα τοπικά δίκτυα και αυτό είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό για τις εταιρείε, κυρίως οι εταιρείε ε, που προσφέρουν υπηρεσίες προς άλλες επιχειρήσεις, ε, προς μικρές βιομηχανικές μονάδες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή ακόμη και στη δημόσια διοίκηση, αλλά και προς την νέα αγορά καταναλωτών. Χρειάζεται η ασφάλεια και για τους καταναλωτές, δηλαδή family όροι ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις και δικαιώματα, family όροι ως προς την πρόσβαση στο διαδίκτυο και προφανώς εφόσον μιλάμε για μία ήπειρο δεν μπορεί να ε, υπάρχει το μεγάλη διακύμανση στις τιμές, ε, να έχουμε εκατονταπλάσια τιμή από, διαφορά τιμής ε, από χώρα σε χώρα. Το ίδιο για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στην Ευρώπη. Ε, το κόστος περιαγωγής ε, από οικονομικής πλευράς δεν αιτιολογείται. Θα ήθελα να ε, μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτά τα τρία σκέλη που παρουσίασα. Πρώτον, ο πρώτος πυλώνας είναι το ενιαίο σύστημα διοδότησης. Τι είναι αυτό, είναι σαν διαβατήριο ένα διαβατήριο που ε, αναγνωρίζουν όλα τα κράτη-μέλη και είναι πολύ περίεργο ε, που επιχειρήσεις τελεπικοινωνιακών υπηρεσιών σήμερα χρειάζονται 28 διαφορετικές άδειες. Ε, το φυσικό θα ήταν να εξασφαλίσουμε ότι η αδειοδότηση που εκδίδεται από το κράτος αυτόματα αναγνωρίζεται από όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά υπάρχουν πιο προηγμένες και περίπλοκες λύσεις, μια κεντρική αρχή που θα αναλάβει τις αδειοδοτήσεις, αλλά αυτό θα μας οδηγήσει σε περισσότερο κεντρική διακυβέρνηση και άρα γραφειοκρατία, αντίθετο προς τους στόχους της πρότασης. Εμείς επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρον την υφιστάμενη διακυβερνητική υποδομή στην ε, Ευρώπη, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές που ασχολούνται με το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων να μπορέσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά. Αυτό δεν δημιουργεί νέα γραφειοκρατία, ούτε ε, νέους κεντρικούς οργανισμούς που κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζονται ε, αυτή τη στιγμή. Ενιαία αδειοδότηση λοιπόν. Πολύ απλή αρχή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εκδίδουν ε, την άδεια προς μία επιχείρηση και μπορεί να λειτουργήσει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εάν το επιθυμεί επιχείρηση δεν υποχρεούται, εάν όμως επιθυμεί να ε, αναπτύξει δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει το σήμα της Ευρωπαϊκής Επιχειρήσης. Πρέπει βεβαίως να δραστηριοποιείται σε τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Και όταν ε, μιλάμε για τα τεχνικά ένδικα μέσα, παραδείγματο χαρή, αν ε, αποκτήσει πολύ μεγάλη θέση στην αγορά σε κάποιο κράτος μέλος αυτή η επιχείρηση, τότε δικαιούται η επιχείρηση να έχει ισότιμη μεταχείριση για τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, όταν είναι ε, συνθήκες θα πρέπει να έχει ισότιμη μεταχείριση. Αυτό κατοχυρώνεται από το ότι ζητήσαμε αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβάλλουμε βέτο σε σχέση με τις δικαιοδοτικές εξουσίες μία χώρα σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα σε σχέση με το ευρωπαϊκό σε εισαγωγικά διαβατήριο. Αν μια επιχείρηση πάει σε ένα κράτος μέλος και χρησιμοποιήσει ε, ρυθμιστικά ένδικα μέσα, τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξασκήσει αυτές τις ορμοδιότητε σε διαβούλευση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Εξυπακούεται για ποιο λόγο, διότι θέλουμε να εγγυηθούμε ότι οι επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα και θέλουν να επιτύχουν μια ε, οικονομία κλίμακας θα πρέπει να έχουν ασφάλεια δικαίου. Να ξεκαθαρίσω όμως ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει ότι η πρόσβαση στα τοπικά δίκτυα πρέπει να ρυθμίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι. Αυτό ε, Βάσει του σχεδίου πρότασής μας ε, θα ρυθμίζεται σε τοπικό επίπεδο και πρόκειται για εγχώριες αποφάσεις ε, των τοπικών ρυθμιστικών αρχών. Όταν υπάρχει επιθυμία δραστηριοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτω ώστε να ισχύουν κάποιοι ενιαίοι εναρμονισμένοι κανόνες. Ε, το, κομμάτι του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, πολύ σημαντικό. για όποιον φορέα και να μιλάμε, για οποιαδήποτε επιχείρηση και να μιλάμε, είναι σημαντικό το ζήτημα. Έχουμε έχουν όλοι ε, την ίδια ενδιαφέρον για το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων. Ε, είναι αρκετά απλό να σας εξηγήσω αυτό το θέμα. Το 6% έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή σε σχέση με το παγκόσμιο φάσμα. Ε, και με όλο το σεβασμό ε, είμαστε όπως ήταν ε, η Αφρική πριν από 40 χρόνια. Για πολλούς λόγους. Αν δείτε τι έγινε μετά την πολύ σημαντική απόφαση του προσδιορισμού του προγράμματος της πολιτικής ραδιοφάσματος, για τα, τις ε, ζώνες 800 MHz και τα λοιπά, ε, όταν έγινε ο καταμερισμός των ραδιοσυχνοτήτων δηλαδή, Ε, είδαμε ότι δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη σε κάποια κράτη-μέλη. 17 μονοκράτη από τα 28 έχουν πάρει το κομμάτι τους από το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι δυσκολίες συνεχίζονται και δεν βλέπουμε το φως στην άκρη του τούνελ προς το παρόν. Αυτό στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών δημιούργησε ιδιαίτερη ανασφάλεια, ανασφάλεια για τις κατασκευαστικές εταιρείες και ως αποτέλεσμα, και είναι λυπηρό που το λέω, ο, η οι ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες δεν έχουν χώρη αγορά, δεν παράγουν εδώ, είναι αλλού στον κόσμο. Γι' αυτό και η ασύρματη Ευρώπη πρέπει για να υλοποιηθεί ε, να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Πώς θα γίνει αυτό, να ενισχύσουμε την ε, διακρατική συνεργασία για τη χορήγηση ε, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση και τοποθετείται εν συνεχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι Ε, η ταχύτητα και το κατά πόσο τα μικροκύτταρα μπορούν να μας οδηγήσουν σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε συνδυασμό με το νέο σύστημα διοδότησης στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα θα δίνεται η ευκαιρία χορήγησης ε, ασύρματων ζωνών χωρίς ε, ε, γραφειοκρατία και χωρίς ε, να υπάρχουν ε, ανεπιθύμητες παρεμβολές λόγω συνοστισμού στο δίκτυο. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσφέρουν υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, προς την δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη οφείλουν να υπάγονται σε έναν αρμονισμό γιατί αλλιώς δεν, μπορεί να, δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πεδίο που δεν είναι ενίο και επίσης οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν ποιοι είναι κανόνες του παιχνιδιού όταν ο στόχος είναι να παράσχουν ε, υπηρεσίες σε μια επιχείρηση ε, που ε, δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας περάσω τώρα στους καταναλωτές. Ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να προσφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά μια διασυνδεδεμένη υπήρου. Πρώτον, συμβατικέ προϋποθέσεις. Εναρμονισμένες συμβατικέ προϋποθέσεις δημιουργούν ασφάλεια για του χρήστες. Οι χρήστες ξέρουν ποια είναι τα δικαιώματά τους όταν θέλουν να αλλάξουν ε, φορέα παροχής υπηρεσιών, ε, γνωρίζουν τα χρονικά περιθώρια, ε, επιτυχάνουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για τα τιμολόγια, ποια είναι η πολιτική τιμών ε, του, του φορέα παροχής. Γι' αυτό και είναι δύσκολο ε, να ε, προσδιορίσουμε με σαφήνεια μια χάρτα δικαιωμάτων των καταναλωτών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Για τους καναλωτές έχουμε επίσης την πρόταση να, να υπάρξει νομοθεσία για τα βασικά χαρακτηριστικά πρόσβασης στο διαδίκτυο. Αυτό βεβαίως έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλουμε υπερβολική γραφειοκρατία ρυθμίσεις. Προτείνουμε νομοθεσία πιο ανοιχτό λοιπόν και διαφανές σύστημα για να υπάρχει λογοδοσία. Νομίζω ότι η πρότασή μας λοιπόν είναι ισορροπημένη. Είναι φυσικά μόνο πρόταση. Τώρα τα δημοκρατικά όργανα θα αποφασίσουν ε, ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Αλλά προσπαθούμε με πολύ διαφανή, ορατό για όλους τρόπο να προχωρήσουμε. Θα θυμάστε, κάναμε συστάσεις και από νομική άποψη θέλουμε να αποφύγουμε ασάφειες και διαφοροποιήσεις στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε την ουδετερότητα του διαδικτύου, άρα προτιμούμε την νομοθεσία. Είναι η πιο προοδευμένη στον κόσμο η νομοθεσία μας σε σχέση με τον Αμερικανικό νόμο για την ουδετερότητα του δικτύου είναι πολύ πιο φιλική προς τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, για χρήστες κινητών στην Αμερική ε, υπό προϋποθέσεις απαγορεύεται ε, η ε, φόρτωση βίντεο, ενώ εμείς δεν το επιτρέπουμε, είναι ανοιχτό το διαδίκτυο και η διαχείριση της κυκλοφορίας στο δίκτυο θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην εμπεριέχει διακρίσεις. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες και αν θέλετε να τις συζητήσουμε. Εδώ στην Επιτροπή σας ή και σε άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ πολύ. Α, μισό λεπτό για την περιαγωγή μια, μια φράση. Ή μερικές. Τι προτείνουμε για την περιαγωγή. Αλλαγή προτύπου. Αλλαγή προτύπου. Αρχή μας όχι επιπλέον κόστος για την περιαγωγή από την 1η Εβδόμου 14. έχει μειωθεί τόσο πολύ το κόστος γενικά για τις εταιρείε, άρα δεν χρειάζεται να πληρώνουν για περιαγωγή περισσότερο. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης, το πρότυπο. Η περιαγωγή είναι τμήμα της οικονομικής δραστηριότητας και φύσης των τηλεπικοινωνιών. Ακόμη και αν περάσει από δίκτυο σε δίκτυο υπάρχει εξωτερικό κόστος. Άρα πρέπει να, να το θεωρήσουμε ως ένα ε, ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο. Άρα το κόστος πρέπει να είναι στοιχείο του τρόπου τιμολόγησης. Θα πρέπει λοιπόν όλοι οι πάροχοι να έχουν το σωστό δίκτυο σχέσεων μεταξύ τους, ούτως ώστε αυτό το κόστος της ε, περιαγωγής να ενταχθεί στον τρόπο υπολογισμού του κόστου, του κόστους τους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι σύντομα θα καταργήσουμε το κόστος περιαγωγής. Αυτό είναι πολύ καλό νέο. Σας ευχαριστούμε πολύ, δόκτωρα Βιόλα, για τα όσα μας είπατε και ξεκινάει η συζήτηση. Γνωρίζετε βεβαίως ότι θα έχουμε και άλλες φορές τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα ε, αυτό. Άλλωστε θα έχουμε και την ευκαιρία όταν θα, παρουσιαστεί, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της μελέτης επιπτώσεων και άλλωστε θα ε, υπάρξει και στις 5 Νοεμβρίου ενδεχομένως ακρόαση με το ίδιο θέμα της Επιτροπής Ήτρε και θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Δεν έχουμε ακόμα ενδείξεις ε, των εισηγητών ε, και των, ε, της εισηγητρίας μάλλον ή των σκιωδών γιατί θα ληφθούν οι αποφάσεις αυτές ίσως και σήμερα το απόγευμα στη συνεδρία των συντονιστών. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Δεκαστήγιο, Μαδουρέλα, Όκμαρ, Τρότμαν, Ρούμπιχ, αυτές, ε, αυτοί οι αγορητές που και ο κύριος Σοντή ε, παρακαλώ πολύ να μην μακρηγορήσετε γιατί θα, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και την απάντηση του δόκτωρου Βιόλα ο οποίος ε, θα πρέπει να φύγει γύρω στις 11 μας το είχε πει από πριν άλλωστε. Pas de problème, pense que Να επιχειρήσουμε όλοι να είμαστε σύντομοι γιατί έχουμε και πολλά άλλα θέματα σήμερα το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που συζητάμε. Ευχαριστώ την Κομισιόν που απάντησε τόσο σύντομα στο αίτημά μα να μα παρουσιάσει το θέμα αυτό. Δεν θα μιλήσω για το περιεχόμενο, αλλά ε, για θέματα διαδικασίες. Ε, δεν θα αναφερθώ στην ε, ιδιαίτερη σημασία που έχει η ανάπτυξη όλων αυτών των στοιχείων σύνδεσης της Ευρώπης για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα ε, σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Για μένα δεν έχει έρθει ακόμη στιγμή. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη συνεδρίασή μας γιατί έχουμε μια πρόκληση ενώπιόν μας Άρα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια και αποφασιστικότητα. Όπως είπε και η Επίτροπος και άλλοι συνάδελφοι και εδώ και αλλού, χτες κάναμε μια συζήτηση με την κυρία Κρούζ στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για το Διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτό που τονίθηκε τονίστηκε είναι ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Αυτό το πακέτο μας υποβάλλεται πολύ αργά. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την ευθύνη μας, την ευθύνη μας να καθορίσουμε μια θέση έχοντας όλα τα στοιχεία που μας επιτρέπουν να το συζητήσουμε, να το σκεφτούμε τεκμηριωμένα. Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια είναι η θέση μου. Διότι... Ποια είναι λοιπόν η θέση μου. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Ρομπέρτο Βιόλα, ότι είναι πακέτο αυτά τα θέματα. Η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο έχουν υποχρέωση να καθορίσουν τη θέση τους σε σχέση με αυτό το πακέτο. Παρά κάποια έλλειψη ε, σύνδεση μεταξύ των στοιχείων, είναι λογικό να τα αντιμετωπίσουμε μαζί. Νομίζω πως θα ήταν σκόπιμο, όχι από τεχνική άποψη βέβαια, γιατί δεν θα είχε έννοια. Πρέπει λοιπόν, δεν θα πρέπει να κάνουμε απλώς ένα κατάλογο θεμάτων, ε, να βάλουμε λίγο από να βάλουμε λίγο από το άλλο. Όχι, δεν προχωράμε έτσι. Πρέπει να έχουμε συνέστηση τι μπορούμε να κάνουμε και ποια είναι τα όρια της δυνατότητας παρέμβασή μας. Πρέπει να έχουμε θέση στην Ολομέλεια. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε, να συμφωνήσουμε στην Ολομέλεια. Δεν είναι θέμα να αναπτύξουμε τη σχέση μας με το Συμβούλιο. Πρέπει να καταλήξουμε σε θέση στην Ολομέλεια. Το Μάρτιο. Με αποτελεσματικότητα με φυσικά το υψηλό επίπεδο εργασίας ε, και υπευθυνότητα που έχουν τα μέλη της Επιτροπής μας και η γραμματεία μας οπωσδήποτε πρέπει οπωσδήποτε αυτό που θα κάνουμε, εάν το κάνουμε έτσι, να έχει δυνατότητες να περάσει μετά, να επιτύχει. Είναι λοιπόν πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόταση της Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, με τη σύνθεση που έχει μετά από πέντε χρόνια καταλήγει, καταλήγει να συζητάει αυτά τα θέματα, άρα πρέπει να ανταποκριθούμε. Και στις συζητήσεις που θα κάνουμε εδώ, στην Επιτροπή μας, να δούμε ποια θέματα θεωρούμε ότι είναι τα πιο σημαντικά και άρα πρέπει να τα τονίσουμε και ποια είναι λιγότερο σημαντικά. Αλλά, συνοψίζοντας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση. Πρέπει ότι μπορεί να την αντιμετωπίσουμε σωστά, έγκαιρα και το σωστό περιεχόμενο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως πακέτο. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί το Συμβούλιο ή κάποια κράτη-μέλη θέλουν να πάρουν λίγο απ' όλα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά η θέση του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι συνεπής. Γιατί το θέμα αυτό είναι κλειδί αν θέλουμε να προχωρήσουμε ή όχι. Τερέσα Μαδουρέλ. Παρακαλώ να κοιτάζετε και το ρολόι. Γιατί καθυστερήσαμε. Θα επιχειρήσω να είμαι σύντομη. Η ομάδα μου συμμερίζεται την ανάλυση της Κομισιόν για την κατάσταση που υπάρχει στον τομέα. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών οπωσδήποτε έχει ανεπάρκειες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου και έχουν πολύ αρνητικέ συνέπειε για του Ευρωπαίου καταναλωτέ όσον αφορά την τιμή, την πρόσβαση σε υπηρεσίε ε, υψηλού επίπεδου όπω ε, μα εξηγήθηκε από τον κύριο Βιόλα, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του στην Επιτροπή μα. Είναι σαφέ ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ευρώπη. Είναι ζωτικό, συμφωνούμε όλοι. Ωστόσο, επίση ισχύει ότι το πακέτο, και εδώ συμφωνώ με την κυρία Δεκαστήγιο, μας υποβάλλεται με πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Αλλά επειδή είναι πολύ ευρύ αυτό το πακέτο, θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε φιλόδοξη συμφωνία πριν το τέλος της θητείας και πιστεύω ότι ορισμένα από τα μέτρα έχουν καθυστερήσει. Ή πολύ νωρί, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, γιατί υπήρξε και η πρόσφατη μεταρρύθμιση κάποιων πλευρών. Φοβόμαστε λοιπόν ότι θα αντιμετωπίσουμε δυσχέρειες, όπως ε, αυτές που αντιμετωπίσαμε στις προηγούμενες προσπάθειες. Όπως είπε ο κύριος Βιόλα για το θέμα της περιαγωγής, είναι πολύ πρόσφατη η τελευταία μεταρρύθμιση της περιαγωγής, για την οποία η ομάδα μου ήταν υπεύθυνη εμείς. Είχαμε τονίσει ότι θα έπρεπε να καταργηθεί το κόστος του, της περιαγωγής. Ε, ελπίζω η θέση κάποιων άλλων ομάδων να αλλάξει και το ίδιο ισχύει για κάποιε προτάσει εναρμόνιση ε, που κάνει η Επιτροπή. Νομίζω ότι ιδίω στο Συμβούλιο θα αντιμετωπίσουν μεγάλε αντιδράσει. Γιατί όπως ξέρετε αυτό παραδοσιακά είναι εθνική αρμοδιότητα. Τα αναφέρω μόνο ως παραδείγματα των ε, συγκρούσεων που μπορεί να μας εμποδίσουν να επιτύχουμε ικανοποιητική συμφωνία. Αλλά τα μέτρα αυτά έχουν τεράστιο δυναμικό να ωφελήσουν τον τομέα, τους καταναλωτές, όπως πολύ καλά ε, εξηγήσατε και βεβαίως και η διανομή ε, συχνοτήτων και ένα ενιαίο σύστημα οπωσδήποτε θα εξασφάλιζε πιο ανοιχτή πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, η ουδετερότητα του διαδικτύου, ε, ένα ανοιχτό διαδίκτυο βεβαίως. Δεν είναι απλώς θετικά για τον καταναλωτή, είναι θεμελιώδη για να υπάρξει πρόοδο στον τομέα των υπηρεσιών. Οπωσδήποτε η ομάδα μου θα το υποστηρίξει. Και βεβαίω ε, καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Και καταλήγω. Θα έλεγα ότι η ομάδα μου. Πολλά θα μπορούσα να πω, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Η ομάδα μου λοιπόν μελετάει την πρόταση σε βάθος, όπως είπε και η Πρόεδρος. Θα ορίσουμε σύντομα τους εισηγητές και σας εγγυώμαι ότι η ομάδα μου θα εργαστεί για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τους καναλωτές, για τον κλάδο, για να έχει ανταγωνιστικότητα, για να συμβάλλει με το τεράστιο δυναμικό που έχει στον εξυγχρονισμό και την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τελείωσαν οι συντονιστές. Ε, περνάμε τώρα στους ε, συναδέλφους ε, Όκμαρ, Thank you very much. Um, Ευχαριστώ. Πολύ καλή ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε όχι μονάχα το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και την ίδια αυτή την πρόκληση. Στα Ηνωμένα Έθνη η Επιτροπή Εβραίου Σπάσματος συζήτησε, την, παρουσίασε την έκθεση του και ε, είπε ότι η τεχνολογία της, του φάσματος ε, για, την, για τα κινητά είναι ε, ιστορικά η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη και βεβαίως δείχνει και το πόσο γρήγορα αλλάζουν και οι συνθήκες και μπορούμε να καταλάβουμε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και στην τηλεπικοινωνίες και στην κοινωνία και στην βιομηχανία. Από αυτή την άποψη άποψη λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν αλλά φυσικά και κυριότερα τις ευκαιρίες. Η Ευρώπη κάποτε ήταν ηγέτιδα όσον αφορά το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες. Η Νόκια ας πούμε ε, είναι ενδεικτικό ότι πούλησε την ε, εταιρεία της ε, στην Microsoft πριν από μερικές εβδομάδες και το κόστος ήταν 130 δις ενώ ξεκίνησε σαν μια μικρή εταιρεία και η Apple κοστίζει 350 δις. αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν οι συνθήκες και από τη δική μας άποψη πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας όχι μόνο στην αύξηση των ικανοτήτων μας, αλλά ε, και την ε, διαμόρφωση του σωστού περιβάλλοντος για την ε, βιομηχανία και τη διαμόρφωση ενός γενικότερου ε, σωστού περιβάλλοντος. Βλέπω ότι στην ανακοίνωσή της η Επιτροπής λέει, βλέπω μάλλον την εικόνα ενός τουρίστα που μιλάει στο κινητό του ξαπλωμένος στη θάλασσα. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό το roaming, η περιαγωγή χρειάζεται όχι μόνο για τον τουρίστα αλλά για την ανάπτυξη των ιδίων των βιομηχανιών μας. Δεν είναι για τον τουρίστα, είναι για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί και θα ξαναπάρει ηγετικό ε, ρόλο και ηγετική θέση η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ήδη από την εφιστάμενη νομοθεσία ε, να δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε και ποιες είναι οι αλλαγές οι οποίες μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε στις τηλεπικοινωνίες. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα ε, γιατί πολύ αργά ήρθε αυτή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από τη δική μας πλευρά εμείς θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις στρατηγικές αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα και πρέπει να είμαστε βεβαίως και ορθολογιστές γιατί Εάν δεν κάνουμε τις ε, αλλαγές που πρέπει γρήγορα, ε, ε, τότε θα, αυτά που χάνουμε εμείς, τα ποσοστά της αγοράς που χάνουμε εμείς, θα τα κερδίσουν κάποια άλλα μέρη του κόσμου. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ευκαιρίες και να δράξουμε και τις ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τρότουμάν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πατρίτσια. Άκουσα αυτήν την εισαγωγή του κύριου Βιόλα, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι, ε, ο οποίος μας είπε ότι δεν πρόκειται εδώ για μια πρόταση έτσι από κομμάτια ατάκτο ερημένα, αλλά είναι ένα πακέτο, είναι μια δέσμη. Ε, εγώ άλλωστε έχω κάνει και μια έκθεση για την Peace Approach και ε, Νομίζω ότι για να πούμε πραγματικά ότι πρόκειται για πακέτο θα πρέπει να απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, Έχουμε δύο αντικρουόμενες λογικές. Από τη μία την ρύθμιση, που είναι η ρύθμιση του ισχύοντος πακέτου Telecom, τηλεπικοινωνιών, το πακέτο του ανταγωνισμού, ε, που αφορά την ε, ολοκλήρωση της αγοράς. Είναι δύο διαφορετικές ε, λογικές και ο κύριος Βιόλα μας λέει ότι εδώ έχουμε ένα ενδιάμεσο βήμα. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τον τρόπο να δούμε εάν αυτό το βήμα είναι ενισχυτικό ε, ή αν αντιθέτως αποτελεί οπισθοδρόμηση και αποδυναμώνει ακόμα περισσότερο τον τομέα. Όσον αφορά το διαβατήριο, ε, λέτε δεν είναι, ίσο, ε, δεν είναι ισότιμο αλλά είναι παρόμοιο. όταν θα πρέπει να ε, ρυθμιστούν ε, ε, οι έννοιες έτσι ώστε να δούμε πότε η Κομισιόν μπορεί να ασκήσει βέτο, τότε αυτό το similar, το παρόμοιο, δεν μας καλύπτει. Ε, εδώ θα πρέπει να, να δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο γιατί διαπιστώνω κύριε Βιόλα ότι και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε σε ένα πρόβλημα επικουρικότητας όταν λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει για τον τομέα ευρωπαϊκή ε, ρύθμιση. Αυτό το σημείωσα με προσοχή. Επομένως δεν, δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς και άλλωστε ε, είδαμε και την αξιολόγηση για τον Μπέρεκ, ε, του Μπέρεκ μάλλον όσον αφορά την πρόταση έτσι όπως την ε, τοποθετείτε σήμερα. Τρίτον, θα ήθελα η Κομισιόν όταν ψηφιστεί ε, το πακέτο τηλεπικοινωνιών. Θα ήθελα λοιπόν να είχε βάσει αυτού του πακέτου ε, κάνει μια γενικότερη βιομηχανική πολιτική. Ε, είδα τι μέτρα έχετε πάρει για τη Vodafone και για κάποιον άλλον επίγειο πάροχο στη Γερμανία. Έχετε κάνει κάτι άλλο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο τι γίνεται σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως. γιατί διαφορετικά διαφορετικά έχουμε διαρκή απώλεια ε, δυνατότητας ε, ε, των επιχειρήσεων και των βιομηχανών μας. Επίσης δεν είδα μια σαφή πρόταση όσον αφορά μια, ένα σταθερό πρόγραμμα για τις οπτικές ίνες στην Ευρώπη και την, το δίκτυό τους και επομένως αυτό δεν είναι σωστό για τους πολίτες. Δεν, δεν είναι μονάχα δεν είναι μονάχα πρόβλημα σε σχέση με το πόσα πληρώνει για το πακέτο που έχει ο καταναλωτής, αλλά και τι ποιότητα έχει και τι δυνατότητα του προσφέρει το πακέτο αυτό. Επομένως, η Κομισιόν θα πρέπει να ε, ε, ε, κάνει ένα, να εκπονήσει ένα πραγματικό συνολικό σχέδιο. Πρέπει να δούμε τι γίνεται και στις χώρες του Νότου και στις χώρες της Ανατολής και του Βορρά, γιατί αυτή η ίδια συνδεσιμότητα θα αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο ανταγωνιστικό ε, και επομένως ε, εδώ ε, το ζήτημα δεν αφορά μονάχα το κόστος και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις του κόστους αλλά είναι ένα πρωταρχικό ζήτημα το οποίο αφορά την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Δεν πρέπει να συζητάμε για στρατηγική μονάχα για την ευρωπαϊκή χαλιβουργία αλλά και για τις ίνες. Και επομένως ε, ε, νομίζω ότι εδώ δεν θα πρέπει οι προσπάθειες που θα καταβληθούν να αφορούν μονάχα την εξέβρεση πόρων ή χρηματοδότησης. Πιστεύω αντιθέτως ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο γενικό πλαίσιο το οποίο δεν το βλέπω τώρα. Όσον αφορά το ε, διαβατήριο. Φοβούμαι η κυρία Βιόλα και θα ήθελα απάντηση από αυτού είναι ότι αυτό το διαβατήριο δεν με βρίσκει αντίθετη, μπορεί να είναι κάτι θετικό, αλλά ε, ε, φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο ε, θα ενισχυθούν μονάχα οι πλούσιοι και μεγάλοι και όχι οι μεσαίου μεγέθους που θέλουν όμως έτσι μια όθηση. Τέλος. Το νέφος ε, είπατε ότι είναι απολύτως απαραίτητο για την, ε, στρατηγική, την ψηφιακή στρατηγική. Γνωρίζετε ότι ε, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε εύκολα να συζητήσουμε, κυρίως στα πλαίσια των συζητήσεων της εταιρική σχέσης ελεύθερων συναλλαγών με, την, με τις ΗΠΑ. Η δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων των Ευρωπαίων είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο. Επ' αυτού λοιπόν και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, θεωρώ ότι η οικονομική ανάλυση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολλέ. ελλείψεις. Ε, το, την αξία των στοιχείων, την αξία των συνδέσεων, την αξία των μετοχών και την αξία τη βιομηχανία. γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ όλοι να καταβάλλετε μια προσπάθεια, έτσι πληρώσουμε στην ώρα μας ε, το θέμα και να έχουμε και την απάντηση του κύριου Βιόλου, ο οποίος πρέπει να φύγει. Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν να μιλήσουν οι επόμενοι, σύντομα να μιλήσουν οι επόμενοι ομιλητές. Έρτσοκ, Ρούπικ, Λάμπερτ, ο Ντι και κλείνει ο κατάλογος των αγοριτών. Χέρτζοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Χαίρομαι που είμαι στη σημερινή ακρόαση, αλλά κύριε Βιόλα, ένα χρόνο νωρίτερα καλό θα ήταν να μας είχατε παρουσιάσει αυτή την πρόταση. Εγώ συμφωνώ με τους συναδελφούς, έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά για τρεις λόγους τουλάχιστον. Έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με τον κόσμο, η αντιπροσωπεία της Ήτρε μόλις ήρθε από την Κορέα. Έχουν 5G δίκτυα, ούτε καν 4G. Καταλαβαίνετε, τρέχει ο κόσμος και εμείς ε, είμαστε πολύ πίσω. Πολύ πίσω επίσης σε σχέση με τις ανάγκες. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να είναι διασυνδεδεμένοι καταναλωτές, οι πολίτες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητάνε την διασύνδεση και άρα έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με τις ε, ε, ανάγκες ε, των Ευρωπαίων διασυνοριακά στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Και κύριε Βιολέ, έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με την νομοθεσία και το νομοθετικό μας πρόγραμμα. Δεν θα κατηγορηθεί ο νομοθέτης αν δεν ολοκληρώσουμε στην πρώτη ανάγνωση. Εγώ είμαι αρμόδια και για άλλους ε, φακέλους και αν για να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου έπρεπε εγώ να έχω φροντίσει, να έχω τελειώσει μέχρι 3 Σεπτεμβρίου για να τηρήσουμε και την προθεσμία για τη μετάφραση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται άοκνα και σκληρά ε, ε, και μετράει κάθε λεπτό καθυστέρηση. Δεν μπορούμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αν δεν προχωρήσετε κι εσείς και εμεί δεν θα υπομιστούμε την ευθύνη για την καθυστέρηση, είναι άδικο ε, και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Τέλος, για το περιεχόμενο το σχολίασαν οι συνάδελφοι, τα έχουν πει όλα. Αλλά επειδή είμαι εισηγήτρια και για άλλα συναφή ζητήματα, θέλω να σα υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε μόνο διασυνοριακό πρόβλημα, έχουμε και στο εσωτερικό πρόβλημα. 30% των Ευρωπαίων πολιτών ε, διαβιούν στην Ευρωπαϊκή Ήπεθρο. Δεν είναι διασυνδεδεμένοι. Διευρύνεται το ψηφιακό χάσμα καθημερινά, νέα μορφή διακριτική μεταχείριση ε, και όσοι ζουν στην Ήπεθρο υφίστανται διακριτική μεταχείριση. Σα παρακαλούμε να περάσετε το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο ώστε ε, αυτό το, για αυτό το συνολικό πακέτο να μην αφήσετε πίσω το άλλο συναφές ε, πακέτο για τις ευρυζωνικές ε, συνδέσεις, γιατί ε, έχετε μεγάλο ρόλο να παίξετε σε αυτή την καθυστέρηση που δημιουργείται. Ο κύριος Ρούμπικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που με ενοχλεί, ότι ενώ είναι τόσο σημαντικός τομέας και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, πολύ σημαντικός, υπάρχει τόση καθυστέρηση, με τόσο ράθιμο ρυθμό δημιουργείται η ενιαία ώρα. Όταν προσπαθώ να κοιτάξω το facebook ή να κάνω κάποιο googling, πληρώνω για κάθε gigabyte 3 ευρώ στο σπίτι μου. Εάν το επιχειρήσω σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, μου κοστίζει 540 ευρώ. Στο σπίτι μου λοιπόν 3 ευρώ, στο δρόμο 540 γίγα. Και αν φύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να κοστίσει μέχρι 14.000 ευρώ. Ένα μπάιτ. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν ε, να είναι αγορά αυτό που να λειτουργεί. Τρία στο σπίτι μου και εκτός 540 ευρώ. Είναι σκάνδαλο. Πού διάολο ζούμε. Τι κατάσταση είναι αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ασκεί περισσότερη πίεση, να μην κάνει περισσότερα τόσο ώστε οι πολίτες να μπορούν να κινούνται στην Ευρώπη χωρίς να έχουν αυτές τις διακρίσεις, αυτήν την εκμετάλλευση για το τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι τεράστιο πρόβλημα. Οι νέοι που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας, οι νέοι που είναι στην αγορά, έχουν τεράστιες δυσχέρειες να πάνε σε κάποια άλλη χώρα και να δημιουργήσουν εκεί την ε, επιχείρησή τους. Εδώ υψώνονται αν τα καταργούνται τα σύνορα. Δεν επιτρέπουμε την ανάπτυξη της μελλοντική αγοράς. Θα πρέπει το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύω ότι εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας, όλες οι ομάδες θα κάνουν το καθήκον τους, πρέπει οπωσδήποτε τα εθνικά συμφέροντα που μας εμποδίζουν που ήδη μας στέλνουν μηνύματα ότι ο, πηγαίνετε πολύ γρήγορα. Το διαδίκτυο κάθε μέρα αυξάνεται, τηλεπικοινωνίες θέλουμε, το κοινοβούλιο ακόμη πριν τις εκλογές πρέπει να αποδείξει ότι μπορούμε να κάνουμε το καθήκον μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ευχαριστούμε ε, για αυτό το, αυτή την παρέμβαση που χειροκροτήθηκε. Λάμπερτ. Σημερίζομαι την, το θυμό του Πολ. Αλλά να πω ότι όταν συζητήσαμε τον κανονισμό περιαγωγή 3, roaming 3, είχαμε, την, είχαμε μια ευκαιρία να χτυπήσουμε μέχρι θανάτου το rolling. Και να πω ότι και οι πράσινοι είχαν την άποψη αυτή, δεν ήταν μόνο οι σοσιαλιστές μπορούσαμε να πούμε να προσθέσουμε δηλαδή στην πρόταση της Κομισιόν ότι πρέπει να σταματήσει το roaming εντελώς και τότε όμως δεν είχαμε την πλειοψηφία. Φαίνεται ότι τώρα και χαίρομαι γι' αυτό υπάρχει αυτή η πλειοψηφία κατά αυτή την έννοια. Αλλά να κάνω και ένα παραλληλισμό με αυτά που κάνουμε ας πούμε στην ΕΚΟΝ ε, προσθέσαμε ε, κάποια στοιχεία στην πρόταση της Κομισιόν όσον αφορά τη διαφάνεια, όσον αφορά ε, την χρηματοδοτική ε, ρύθμιση και θεωρώ ότι η Επίτροπος Κρούσα δεν ήταν στο πλευρό μας όταν χρειαζόμαστε. Τώρα φαίνεται να είναι. Εν πάση περιπτώσει ελπίζω ότι κάτι θα γίνει, αλλά λαμβάνοντα υπόψη το, τις ημερολογικές έτσι, δεσμεύσεις, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ γιατί είσαστε και σύντομος και περιεκτικός. Ο κύριος Οντή παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, πρόσβαση στις υπηρεσίες. Άκουσα τους συναδέλφους ε, να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την ισότιμη μεταχείριση των Ευρωπαίων πολιτών οπουδήποτε και αν ζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο εθίγει αρκετά, έχει συζητηθεί αρκετά. Εγώ άλλωστε εκλέγομαι στην Ήπεθρο ε, και ε, δεν έχουν ακόμα την εντύπωση ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους κακομεταχειρίζονται, αλλά θα έρθει και αυτό και σύντομα μάλιστα. Ε, έχουν την ίδια εντύπωση τουλάχιστον για το εθνικό επίπεδο. Θα ήθελα να μου πει η Κομισιόν γιατί παρά τις αναφορές του, επανειλημμένες αναφορές του Κοινοβουλίου, γιατί δεν αντιμετώπισαν με ισότιμο τρόπο όλη την ενωσιακή επικράτεια. Είπατε ότι δεν δεν υπάρχει δημόσια χρηματοδότηση, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές προσπάθειες κάναμε έτσι ώστε να υπάρχει ε, μια ρεαλίτρια πολιτική αναθεώρηση μετά τις εκλογές. Ε, γι' αυτό λοιπόν μην προδικάζετε το αποτέλεσμα των εκλογών και το τι θα αποτελέσουν, τι θα αποφασίσουν συγγνώμη, οι πολίτες ε, και στη διάρκεια βεβαίως της προεκλογής εξετατείας οπωσδήποτε θα υπάρξει συζήτηση για την ισότιμη μεταχείριση των πολιτών. Εγώ έκανα μία πρόταση ε, που θα, ε, για την ίδρυση ενός ταμείου ε, που θα παίρνει χρήματα μέσα από μία πάρα πολύ μικρή συνεισφορά από τους ίδιους πόρους. Θα πρέπει οπωσδήποτε να εξευρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο πρόσβασης στην ευρυζωνικότητα. Δεύτερον, το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών ε, ε, τηλεπικοινωνιών. Ναι, εγώ θα ήθελα να δω ε, με ποιο τρόπο μεταχειριζόμαστε τους ξένους πάροχους. Υπάρχει μια αρχή η οποία φαίνεται ότι βρίσκει την πολιτική συμφωνία της πλειοψηφίας στο Κοινοβούλιο, δηλαδή την αρχή της αμοιβαιότητας. Εάν δεχτούμε ε, την συμφωνία αυτή, ε, τότε θα πρέπει να δούμε τις ποιες εταιρείες είναι εγκαταστημένες στην Ευρώπη. Η Google, ας πούμε, η οποία ε, μπορεί να έχει μια θεατρική στην Αυστρία, μπορεί να θεωρηθεί ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής ψηφιακού περιεχομένου και επομένως να έχει αυτό το διαβατήριο και λαμβάνοντας υπόψη τα διακυβεύματα θα μπορεί μια ευρωπαϊκή εταιρεία να κάνει το ίδιο πράγμα α πούμε στι ΗΠΑ, Πολιτείε, ε, θα πρέπει πριν υπογράψουμε οτιδήποτε και πριν δεχτούμε ξένε εταιρείε ε, στην ενωσιακή επικράτεια να έχουμε τη διασφάλιση ότι μπορούν να εγκατασταθούν και δικέ μα εταιρείε, αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι αυτή η αρχή τη ε, αμοιβαιότητα ισχύει εάν δεν την έχει συμπεριλάβει την αρχή αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να σημειωθεί και αυτό από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ πολύ. Τσίτσεστερ και Νίμπρε. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε διαβούλευση για αυτό το ζήτημα. Ε, όταν σπέβδουμε έτσι για να νομοθετούμε, έχουμε όλο το χρόνο μετά για να το μετανιώσουμε. Άγγελα Νίμπλε. Ευχαριστώ. Υποστηρίζω όλα όσα είπα συνάδελφοι ότι η πρόταση έχει καθυστερήσει πολύ. Θα ήθελα απλώς να αποστείλω ένα μήνυμα. Όταν ε, μας στέλνετε τόσο αργά στο τέλος της θητείας ένα τέτοιο πακέτο και θέλετε ε, να υπάρχει ισχυρό πολιτικό μήνυμα τότε πρέπει να προωθήσει πολύ το θέμα αυτό η Κομισιόν. Χαίρομαι που είστε εδώ ε, κύριε Βιόλα, αλλά αφού είναι τόσο σημαντικό και θέλετε τόσο πολύ να το προωθήσετε, γιατί δεν είναι εδώ η Επίτροπος. Έξι μήνες πριν από, την, ε, από το τέλος της θητείας θέλετε να μας απασχολήσει. Θα περίμενα ότι θα έπρεπε να είναι παρούσα προσωπικά και η Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Γιακυμαβίτσιους ε, από το Συμβούλιο. Παρακαλώ πολύ να είσαστε πολύ σύντομος και να αναφερθείτε μονάχα σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο στη συζήτηση αυτή και μετά να δώσω το λόγο στον ε, ε, δόκτορα Βιόλα, ο οποίος την αναλάβει και τη δέσμευση να επιστρέψει, γιατί δεν θα μπορέσει νομίζω να απαντήσει με σωστό τρόπο στις ερωτήσεις που του ετέθησαν. Παρακαλώ το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Δ. Βιόλα για την παρουσία του Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Βιόλα για την παρουσίαση που έκανε εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, σαν ε, Προεδρεύουσα έχουμε βεβαίω μελετήσει ενδελεχώς το θέμα και στην Κορεπέρα και στο Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι ένα περίπλοκο και ιδιάζον ζήτημα συμφωνήσαμε, συμφωνούμε με πολλούς από τους παρεμβαίνοντες ε, βουλευτές, ε, δηλαδή ότι ε, δεν ήρθε την κατάλληλη χρονική στιγμή αυτή η πρόταση και, και η πρώτη ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη-μέλη μας δείχνει ότι θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να προχωρήσουμε με το θέμα αυτό. Το χρονικό πλαίσιο είναι ζωτική σημασίας. προσπαθήσουμε βεβαίως να προχωρήσουμε το φάκελο αυτό, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε με βιασύνη και δεν θα μπορέσουμε ίσως να μελετήσουμε ενδελεχώς όλα αυτά τα πολύ ζητήμα, ε, όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα have a debate. Ε, τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο θα είναι εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη ε, και το θέμα αυτό. Θα γίνει μια συζήτηση και ελπίζω ότι θα συμβάλλει ε, στη γενικότερη συζήτηση και θα δώσει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε ενδεχομένως να προχωρήσουμε με το φάκελο αυτό. η φάση εδώ είναι αρχική ε, και σε αυτή την αρχική φάση δεν νομίζω ότι μπορώ να σχολιάσω κάτι παραπάνω ούτε μπορώ να προδικάσω την ενδεχόμενη έκβαση των συζητήσεων. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ξεκινήσουμε την ανάλυση και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε όταν θα έχουμε τις θέσεις και των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι αυτό που θα μπορούσατε να πείτε κι εσείς. Ε, μαζί θα παρακολουθήσουμε την συζήτηση. Πριν ε, δώσω το λόγο στον δόκτωρα Διόλα, απαντώντας και στην ερώτηση της κυρίας ε, Νίμπλερ, η κυρία Κρούς ήρθε στο Στρασβούργο, θα το θυμάστε φαντάζομαι, ε, και έστω και ατύπως παρουσίασε αυτό το, αυτή τη δέσμη. Βεβαίως θα ξαναέρθει στην Επιτροπή μας ε, σήμερα. Εμείς ζητήσαμε και καλέσαμε τον κύριο Βιόλα να έρθει εδώ ε, για να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Γιατί κατά την άποψή μου πριν από την πολιτική παρουσίαση πρέπει να έχουμε και την τεχνική παρουσίαση, να με τι τεχνικέ λεπτομέρειε, αλλά βεβαίω θα έχουμε αργότερα συνάντηση και με την ε, Επίτροπο. Σε 6-7 λεπτάκια λοιπόν, δόκτωρα Βιόλα, μπορείτε να ε, απαντήσετε. Μία πρώτη απάντηση βεβαίω, και μετά βεβαίω θα σας ζητήσουμε να είστε παρόν ε, είτε στην ακρόαση που θα κάνουμε είτε και πιο πριν θα το συζητήσουμε αυτό και στους συντονιστές, ε, γιατί τα ερωτήματα τα οποία υπευλήθησαν είναι ιδιαίτερα σημαντικά και πρέπει οπωσδήποτε να απαντηθούν δεόντως. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Chair, also. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου προσφέρετε την ευκαιρία να επανέλθω, να επιστρέψω εδώ και να απαντήσω λεπτομερώς στα ερωτήματα τα οποία θα καταγράψω με σχολαστικότητα γιατί θέλω να δώσω απαντήσεις σε όλες τις, τις ερωτήσεις. Συγχωρέστε με, θα δώσω τώρα μια γενικόλογη απάντηση λόγω έλλειψη χρόνου. Σας ευχαριστώ για τη νέα πρόσκληση και ευχαριστώ που διευκρινίσατε ότι η Αντιπρόεδρος Νέλη είναι στη διάθεση της Επιτροπής Ήτρε. Μπορείτε να την καλέσετε όποτε κρίνετε απαραίτητη παρουσία σας. Εγώ ε, είμαι εδώ για να κάνω μόνο την τεχνική παρουσίαση. Ευχαριστώ τους ε, συντονιστές για τις φιλοφρονήσεις, για το χρονοδιάγραμμα. Ε, δεν, είναι, ε, δεν εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτε να το διανοηθούμε, να επιβάλλουμε, να ζητήσουμε χρόνο έγκρισης, ε, δεν μπορούμε. Αυτό επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των υπολείπων θεσμικών οργάνων, των δύο συνομοθετών συγκεκριμένα. Αυτό μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσφέρουν υποστήριξη, τεχνογνωσία, ε, να αποκριθούν σε αίτημα τεχνικής ενημέρωσης σε οποιαδήποτε στιγμή, γιατί θα έχουμε ομάδα σε επιφυλακή. Συν το χρόνο νομίζω θα βελτιωθεί η κατάσταση, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα ήθελα όμως Προ το παρόν να υπογραμμίσω κάτι που τόνισαν και τα μέλη της Επιτροπής. Ε, αλλάζει με το ρυθμό, με την, ε, το ρυθμό της ταχύτητας του φωτός ε, ο τομέας. Πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε με πολύ διαφορετικό τρόπο. Καταρχάς, δεν ήταν οι ίδιες ανάγκες που έχουν όλοι οι πολίτες σήμερα σε οποιοδήποτε σημείο της Υπήρου να θέλουν ε, διασύνδεση μέσω κινητού τηλεφώνου υπολογιστή. Εάν διαβάσετε την αξιολόγηση αντικτύπου θα διαπιστώσετε ότι ο μοναδικός στόχος είναι η διασυνδεδεμένη Ευρώπη. Η κατάργηση της περιαγωγής είναι ένα θέμα που, σας, που μας ενδιαφέρει όλους. Δεν είναι μόνο για όσους κάνουν ε, διακοπές ή έχουν ε, ε, μετικήσει σε άλλη χώρα. Για φανταστείτε όταν διασχίσετε τα σύνορα και δεν λειτουργεί πλέον ε, το GPS. Ε, φανταστείτε να μην λειτουργεί το κινητό σας. Ε, δεν μπορούμε να καταργήσουμε το roaming. Η περιαγωγή είναι στη βάση της διασυνδεσιμότητας, οπότε... Δεν είναι ότι εμείς δεν μας αρέσουν διακοπές και δεν πάμε, σε, δεν πάμε διακοπές, αλλά αναγνωρίζουμε τη σημασία που έχει αυτό στην καθημερινή ζωή. Uh, ε, θα πάω στη Ρήγα για να ε, συναντηθούμε με τις ρυθμιστικές αρχές και να καταλάβουμε αν έχουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις, θα τις καταγράψουμε και ο συνομοθέτης αλλά και εμείς θα ακούσουμε με προσοχή τις επιθυμίες τους. Η αντίδραση των αγορών ήταν μάλλον θετική. Ε, μετά το πακέτο τηλεπικοινωνιών και την κοινοποίηση για την αύξηση ε, του 3% θα δείτε ότι όλες οι οικονομικές αναλύσεις είναι θετικές. Βεβαίως, αυτό που δεν αρέσει στους οικονομικούς αναλυτές είναι το κομμάτι των ε, καταναλωτών. Δεν είναι όμως υπεραγορά εδώ, είναι ένα πακέτο μέτρων που πρέπει να γίνει δεκτό ακέραιο. Η πρόταση για την περιαγωγή είναι λογική. Το κόστος των διεθνών κλήσεων δεν είναι σοβαρό πρόβλημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ε, το να τηλεφώνει κανείς από τη Ρώμη στο Βίλνιος που είναι, ε, υπερβαίνει το 1 ευρώ. Ε, αυτό που είπατε για το κατέβασμα δεδομένων από το διαδίκτυο ισχύει και για τις τηλεφωνικές κλήσεις. Είναι απαράδεκτο αυτό το υψηλό κόστος. Είναι πολύ σημαντικό και έχει και ιδιαίτερη συμβολική σημασία να κάνουμε τη διαφοροποίηση ανάμεσα σε μία συνδεδεμένη και μία αποσυνδεδεμένη ήπειρο. Τώρα η σχέση με τις ε, δημόσιες πολιτικές, ε, κυρίως ως προς τη χρηματοδότηση. Αν με ξανακαλέσετε θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ στην αρχή σας μίλησα για τα 8 δις ε, για το rollout και την καινοτόμο χρηματοδότηση. Δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χρηστά τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων και ε, ούτως ή άλλως αυτό συνιστά ήδη προτεραιότητα για τα διαρθρωτικά ταμεία αλλά για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών το βασικό βάρος θα βαρύνει το, τις επιχειρήσεις. Ως προς τη διαβούλευση, έγινε εκτενής διαβούλευση τα τελευταία δύο χρόνια για κάποια από τα τμήματα ε, αυτής της πρώτης, αυτού του πακέτου. Όχι ότι θα έπρεπε να μας ξαφνιάζει αυτό. Όταν άρχισα να δουλεύω σε αυτό το τομέα και τότε δεν είχα πρεσβειοποία, ε, από τότε ασχολιόμασταν με τις αδειοδοτήσεις. Έχουν γίνει έκτοτε 7 διαβουλεύσεις σε πολυάριθμες ομάδες ε, εργασίας. Ε, διαβούλευση από τον Μπέρεκ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μελέτες. Είναι δίκαιο ε, να πούμε ότι δεν έγινε λεπτομερής διαβούλευση για το συνολικό πακέτο, αλλά για όλα τα επιμέρους μέρη έχουν γίνει εκτενείς διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς. Για τον Μπέρεκ έχω την πτήση μου για τη Ρήγα, αυτό σας ευχαριστώ που κάνατε νέες ρυθμίσεις, θα με ξανακαλέσετε για να ξανασυζητήσουμε τα σχόλιά σας για την πρόταση. Μόνο κάτι τελευταίο Πέρα από τη δυνατότητα του Μπέρεκε να επέμβει ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ε, η σημασία του Μπέρεκε έγινε και στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ο ρόλος είναι καταλητικός για την εσωτερική αγορά και για την ανάπτυξη της νέας αγοράς. Θα απαντήσω διεξοδικότερα για αυτό το σημείο στην επόμενη συνεδρίαση και θα προσπαθήσω να διασκεδάσω οποιασδήποτε ανησυχίε. Ζητώ και πάλι συγγνώμη που δεν απαντώ σε όλα τα ερωτήματα τώρα, αν να πω και κάτι τελευταίο για την ε, ολοκλήρωση. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τους κανόνες περί ανταγωνισμού μέσα από αυτή την πρόταση. Οι παίκτες της αγοράς θα αποφασίσουν αν θέλουν ή όχι να επενδύσουν σε άλλες χώρες. Εάν το επιθυμούν, ευπρόσδεκτο είναι και ένα καλό σημάδι για την Ευρώπη, για το μέλλον, αλλά δεν μπορεί κανείς να εξαναγκάσει η ιδιωτική εταιρεία να επενδύσει ε, σε οποιαδήποτε χώρα. Τι γίνεται όμως. Με αυτή την πρόταση δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ε, συρρήκνωση της γραφειοκρατίας. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ε, για την ε, ευχερή χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων με συναφή τρόπο σε όλη την Ήπειρο. Επίσης δημιουργούμε ισότιμες προϋποθέσεις για τις ευρυζωνικές. Εάν τώρα μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για τον, ανταγωνισμό σε τοπικό επίπεδο δημιουργούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις και φυσικά είναι εφαρμοστέ η συνθήκη για τις συνθήκες περί ανταγωνισμού αλλά σε τοπικό επίπεδο μπορούν να γίνουν πλέον όλες αυτές οι κινήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Βιόλα. Ε, ναι, καταλαβαίνουμε ότι έχετε μια δέσμευση χρόνου. Ε, έστω και αυτές οι πρώτες απαντήσεις που μας δώσατε καλές είναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε περαιτέρω γιατί βεβαίως μας απασχολεί εδώ στην Επιτροπή μας. Θα έχουμε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης επιπτώσεων, ε, θα έχουμε την ακρόαση. Ε, όλα αυτά θα αποφασιστούν στους συντονιστές σήμερα το απόγευμα. Θα έχουμε πολλές ευκαιρίες. Ευχαριστώ και την Λιθουανική Προεδρία. Ευχαριστώ σε όσους πήραν το λόγο. Περνάμε στο επόμενο θέμα. θα δώσω τον λόγο αμέσως στον συνάδελφο Μπέντσεν για την έκθεσή του «Αποκάλυψη πληροφοριών με οικονομικής φύσεως και πληροφοριών σχετικά με την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους». Έχουμε στη διάθεσή μας περίπου 30 λεπτά. Ε, ε, να σεβαστούμε λοιπόν όλοι το χρόνο μας γιατί και ο συνάδελφος έχει ε, μετά μια υποχρέωση και πρέπει να φύγει. Ο συνάδελφος Μπέντσεν. Ευχαριστώ. κυρία Πρόεδρε. Ε, η ε, ανάπτυξη των επιχειρήσεων αλλά και ο σεβασμός των υποχρεώσεων δεν είναι δύο ε, αντικρουόμενα ζητήματα. Μπορεί κανείς να έχει εταιρείες οι οποίες αναπτύσσονται καλά και οι οποίες αντιμετωπίζουν και τις κοινωνικές προκλήσεις με τρόπο σωστό. Η πρόταση της Επιτροπής αφορά τον τρόπο με τον οποίο να δίνουν πληροφορίες οι ε, εταιρείε ε, σχετικά ε, με τις πληροφορίες οι οποίες λέω δεν είναι οικονομικής φύσεως όμως που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές για, την, για τους μετόχους σε γενικέ γραμμέ πρέπει να πω ότι με ικανοποιεί η πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, και ε, ε, επομένω το θέμα αυτό του ΕΚΕ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό λοιπόν οι μέτοχοι να ξέρουν τι δραστηριότητε ΕΚΕ και να μπορούν να τι κοινοποιούν εάν στόχος είναι η αύξηση της ε, ε, διαφάνειας, και της δυνατότητας που έχουν ε, οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι μέτοχοι να συγκρίνουν, τότε θα πρέπει να υπάρχει όντως ένα, ένα κοινό πλαίσιο για την αναφορά αυτών των πληροφοριών. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα ε, όπου ε, αυτή η αναφορά της κοινωνικής ευθύνης είναι ε, πολύ συνηθισμένη και μάλιστα είχε καλά αποτελέσματα. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρχουν, να υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης πληροφοριών μη οικονομικής φύσης. Η δικιά μας εμπειρία δείχνει ότι πολλές είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν έχουν ε, αποφασίσει να εμπλακούν στη διαδικασία της ΕΚΕ. Ε, χωρίς να ε, ε, προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτήν την υποχρέωση και μάλιστα το γεγονός της μη εμπλοκής διαδικασία και από πλευράς επιχειρήσεων αποτέλεσε και αποτελεί κακή, κακή φήμη ας πούμε για την εταιρεία αυτή. Θα πρέπει ε, να επιλέξουμε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι ε, σωστό και συμπληρωματικό ε, όσον αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει αυτή η εμπλοκή στη διαδικασία της και να είναι παραγωγική και να βοηθάει τις εταιρείες έτσι ώστε να μπορούν να αναφέρονται σε στοιχεία τα οποία να είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν για κάθε κλάδο ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες, είναι σχετικές με τις δραστηριότητες της εταιρείας και να μην χρειάζεται να αναφέρονται σε μια σειρά θεμάτων άσχετων με τις δραστηριότητες τους. Ευχαριστώ πολύ. Λάγκε, Κρότσμαν, Λάμπερτς. Οι τρεις συνάδελφοι που έχουν εγγραφεί. Ευχαριστώ δυστυχώ. Η σκιώδη συγγήτριά μα δεν είναι παρούσα, δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Γι' αυτό θα αναφέρω μερικά σημεία, αλλά και μερικά δικά μου. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή σας. Βλέπω ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Είναι σημαντικό γιατί ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές αξίες και γι' αυτό το υποστηρίζουμε. Και Πρόσφατα είχαμε τη συζήτηση για την, εργασία, την παιδική εργασία στο Ουσμπεκιστάν ή για τα ατυχήματα στο Μπαγκλαντές. Αυτό καταδεικνύει ότι η συμπεριφορά των ευρωπαϊκών εταιριών και ε, σε σχέση με τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται σε τρίτες χώρες πρέπει να είναι σωστή. Αυτή λοιπόν η εθελοντική συμμόρφωση για κοινωνικά και περιβαλλοντικά στάνταρ πρέπει να προωθηθεί. Είναι λοιπόν σωστή η προσέγγιση μας. Επίσης υποστηρίζω την ε, προσπάθεια να καθορίσουμε ορισμένα σημεία με βάση τα οποία θα πρέπει να κάνουν ε, τις εκθέσεις τους οι εταιρείε. Δεν πρέπει να διαλέγει δηλαδή ο καθένας ποια σημεία θα αναφέρει, ποια κριτήρια, ποιες παραμέτρους θα αναφέρει. Είναι σωστό να υπάρχουν ορισμένες ελάχιστες προδιαγραφές. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν προδιαγραφές και υποστηρίζω την προσέγγιση ε, των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΣΑ του 2011 που πηγαίνει πιο μακριά από οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση Αυτές θα πρέπει να είναι οι προδιαγραφές. Αλλά φυσικά ε, κάποιες επιχειρήσεις υιοθετούν ε, άλλες παραμέτρους και γι' αυτό υποστηρίζω την τροπολογία 5. Να φύγουν αυτές οι εθνικές προσεγγίσεις. Υπάρχουν θεμελιώδη ζητήματα, κοινωνικές προδιαγραφές, περιβαλλοντικές προδιαγραφές. ισότιμη μεταχείριση των φύλων, ε, κοινωνικός διάλογος, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι θεμελιώδη και πρέπει να περιέχονται. Και το θέμα όλων των υπεργολάβων και όλων αυτών των προμηθευτών. Βεβαίως ξέρετε ότι πολύ συχνά στις ε, μεγάλες εταιρείες, πολύ συχνά δεν παράγουν σχεδόν τίποτα. Απλώς αγοράζουν ε, και μετά πουλούν, πουλούν προϊόντα. Άρα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες εργασίας σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Πού διαφωνούμε. Στην τροπολογία 4. Και την 8. Πιστεύω ότι όταν μια επιχείρηση δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της, δεν σέβεται αυτές τις προδιαγραφές, πρέπει να μας εξηγεί γιατί δεν το κάνει. Έχουμε 42.000 επιχειρήσεις. που μας εξηγούν τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Θα ήθελα λοιπόν όσοι δεν θεωρούν ότι πρέπει να το κάνουν να υποχρεωθούν να μας εξηγήσουν γιατί δεν είναι σε θέση να κάνουν αυτές τις εκθέσεις. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η τροπολογία 4, γιατί θεωρούμε ότι όλοι όσοι με βάση αυτή την οδηγία ε, υποχρεούνται να υποβάλουν τέτοιες εκθέσεις θα πρέπει και να το κάνουν. Και έτσι αντιμετωπίζω κριτικά και την τροπολογία 8. Εκεί που συμφωνώ μαζί σας είναι ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται με τον λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο να επιβαρύνουν όσο το δυνατόν λιγότερο τις επιχειρήσεις. Να δούμε δηλαδή από τη μία τι πρέπει να περιέχουν οι εκθέσεις και μετά να δούμε πώς μπορούν αυτές οι εκθέσεις να συνταχθούν με το λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο. Θα συμφωνούσα να τους υποχρεώσουμε λοιπόν σαφείς ε, προδιαγραφές αλλά απλός τρόπος υλοποίησή τους. Ευχαριστώ πολύ. Κρότσμαν. Βεβαίως, ε, κάθε μέρα μιλάμε για την εγγραφή και όλες οι διαδικασίες ε, ε, λέμε ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι απλούστερες. Όταν η Κομισιόν μας λέει πως το κάνουν 2.500 επιχειρήσει αυτές τις προσπάθειες προπάγανδας, εγώ έχω κάνει εκθέσει πολλέ για θέματα αυτά. Τι σημαίνει πρέπει σε όλες τις θηγατρικές εταιρείε να ζητήσετε να σας κάνουν αυτά που θέλετε. Θα πρέπει να αλλάξουν όλες τα συστήματά τους. Πρέπει δηλαδή να πάρουν όλες τις πληροφορίες και να τις βάλουν ε, σε, όλα τα, σε, όλους τους, ε, ε, σε όλα τα συστήματα καταγραφής των δεδομένων τους. Αυτό σημαίνει τρομερές δαπάνες Εάν γίνει μια μικρή αλλαγή σε οτιδήποτε πρέπει όλα αυτά να δούνε, εάν προσαρμόζονται με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες πρέπει όλα αυτά να δούνε ένα συμβατά. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Πρόκειται για τεράστια ποσά. Μπορούμε να τα κάνουμε. Όσοι το έκαναν, το κάνουν μόνο και μόνο για να δείξουν τι καλά σέβονται το περιβάλλον. Βεβαίω υπάρχουν μικρέ ε, χημικέ εταιρείε που το κάνουν, αλλά ξέρετε τι σημαίνει για μια μεγάλη εταιρεία όπω η BASF. Πρέπει λοιπόν να πω ότι εθελοντικά βεβαίω, σωστό, αλλά αν θέλουμε 42.000 επιχειρήσει να τι υποχρεώσουμε και πρέπει να ελέγξουμε αν γίνεται και σωστά. να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ζητάμε και αν με αυτόν τον τρόπο θα επηρεάσουμε θετικά ή αρνητικά την ανταγωνιστικότητα. Και το πρόβλημα που με απασχολεί είναι το επόμενο βήμα. Οι μεγάλες εταιρείε το κάνουν. Το κάνουν. Α, το επόμενο βήμα είναι θα πρέπει να το κάνουν μετά και μικρότερες επιχειρήσεις. Είμαι απόλυτα αρνητικός. Γιατί έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα των ε, εταιρεών αυτά που προτείνει ίσως ένα βαθμό δεκτά ο συνάδελφος Μπένσεν, αλλά γιατί να επιβαρύνουμε επιπλέον τις επιχειρήσεις. Ήδη έχουν τόσο πολλά να κάνουν. 42.000 επιχειρήσεις επιπλέον. Για τις μεγάλες, τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις έχουν επαρκές προσωπικό για να το κάνουν. Έχουν τα ε, συστήματα υπολογιστών και λογισμικών, είναι τόσο μεγάλοι, μπορούν να το κάνουν. Εντάξει, 30.000 30 παραπάνω κόστος δεν τις πειράζει τόσο πολύ. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε και να σκεφτούμε. Κάθε μέρα καλούμε την Κομισιόν ε, ε, να μας κάνει προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας. Αλλά κάθε μέρα υποβάλλονται και νέες προτάσεις νομοθετημάτων που θέλουμε να μας κάνετε και αυτό, θέλετε να μας κάνετε και το άλλο, και θέλουμε να μας αποδείξετε ότι υπάρχει αρκετή, αρκετός σεβασμός για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες, τι εθνικότητα. Χθε ήμασταν σε μια εκδήλωση και μας είπε μια μεγάλη επιχείρηση ότι βεβαίως τα κάνουμε. Εμείς ούτω, ή άλλως θέλουμε τους καλύτερους, δεν μας ενδιαφέρει το φίλο τους, δεν μας ενδιαφέρει η εθνικότητά τους. Πρέπει να μας εξηγήσουν όμως γιατί το κάνουν. δεν είναι δυνατόν να ζητάμε να κάνουν περισσότερα. Πρέπει η Κομισιόν να έχει μια λογική πολιτική. Δεν είναι δυνατόν τη μία μέρα να μας λέει απλούστευση και την άλλη μέρα να τα περιπλέκει τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Λάμπερτ, κύριε Κρότσμαν, πολύ χαίρομαι που βλέπω κάποιον που υπεραμείνεται των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας εμπειρία, αλλά εγώ 22 ε, χρόνια δούλευα στον ιδιωτικό τομέα. Ε, επομένως, εσείς μπορείτε να τα ξέρετε απ' έξω, εγώ τα ξέρω από μέσα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνουν οι μεγάλες εταιρείε. Το να λέει κανεί κάποιος ότι ε, δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε δεσμεύσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί θα πρέπει μετά να το κάνουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αυτό είναι απαράδεκτο. Και εγώ πια έχω βαρεθεί να ακούω αυτή τη φιλελεύθερη αφήγηση ε, να μα λένε ότι ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει είναι αυτέ που κάνουν την κοινοτομία, είναι αυτέ που προχωρούν την οικονομία. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να τις, να τις στηρίξουμε και όταν πρέπει να πάρουμε συγκεκριμένα μέρη, συγγνώμη, αποφάσεις, τότε εμείς οι πράσινοι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι τελικά θέλουμε να πάρουμε πάρουμε συγκεκριμένα μέτρα και λέμε παρακαλούμε βοηθήστε μας να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει. Συμφωνώ απολύτω ότι δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικό το άχθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά αυτές τις ε, ε, επιπλέον εκθέσεις. Θα συμφωνήσω με αυτό. Και επίσης αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν ε, την ικανότητα, δεν έχουν όλους αυτούς τους πόρους που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε αυτήν την υποχρέωση. Ναι, μπορούμε να έχουμε πιο απλή αλλά πιο αποτελεσματική νομοθεσία, αλλά παρόλα αυτά ε, έχω βαρεθεί πια να ακούω και τις μεγάλες επιχειρήσεις να τις βλέπω να παίζουν ε, με τον, με τον νόμο, ε, να παρακάμπτουν τον νόμο, να σκοτώνουν στην ουσία, να είναι υπεύθυνοι για το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στο Πακιστάν και να μην μπορούμε να τους επιβάλλουμε υποχρεωτικούς δεσμευτικούς κανόνες. Ε, στο θέμα των, της αναφοράς των, ε, της αποκάλυψης πληροφοριών οικονομικής φύσεως εμείς κάναμε, ε, πήραμε αποφάσεις όσον αφορά την υποχρέωση που πρέπει να έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να το κάνουμε και εδώ πρέπει να σας πω ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις, το ξέρω πάρα πολύ καλά, το ξέρω και από μέσα, ότι έχουν όλες τις ε, δυνατότητες, ε, γιατί έχουν την, ε, τις δυνατότητες να στηρίξουν αυτό το σύστημα αναφοράς, όπως έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τους μετόχους ψηλά μερίσματα κτλ. Ε, οι μεγάλες, στις μεγάλες εταιρείες θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναφορά και η αποκάλυψη πληροφοριών ε, γενικής ε, φύσεως και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε και δυνατότητα συγκρίσεων. Πρέπει να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία τα οποία δίνουν ε, Βεβαίω μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή την υποχρέωση ε, με ε, δεσμευτικού κανόνες όσον αφορά το περιβάλλον της και την κοινωνική ευθύνη κτλ. Δηλαδή, εάν έχουμε κάποιο τρόπο να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις με δεσμευτικά μέτρα να, να, να ακολουθήσουν τις αρχές του Διεθνου Γραφείου Εργασία, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά δεν γίνεται ούτε αυτό. Και κάτι άλλο ήθελα να αναφέρω, το οποίο αφορά ε, την ανακοίνωση Επιτροπής. Θα θυμάστε ότι όταν συζητήσαμε ε, την ε, αποκάλυψη οικονομικών πληροφοριών είπαμε ότι θα γίνεται αναχώρα ε, και αυτό αποτέλεσε έτσι μεγάλη συζήτηση ε, και η Κομισιόν το αρνήθηκε όταν το ζήτησε το Κοινοβούλιο. Ε, τώρα θα πρέπει να δούμε και τα, τα κατόφυλλα. Ποια είναι τα ελάχιστα, ή τα ελάχιστα μεγέθη. Το κατόφυλλο των μικρομεσαίων επί δύο. Έχω κι εγώ μια σχετική ευελιξία όσον αφορά το θέμα αυτό. Ε, ο Επίτροπος Μπαρνιέ είπε, βασιζόμενος και στη θέση του Συμβουλίου, ότι η αποκάλυψη πληροφοριών μη οικονομικής ε, φύσεως ε, θα, είναι, το, θα, θα αφορά την ανακράτος πληροφόρηση. Ξέρουμε από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου ότι στην ουσία μάλλον αυτό θα το δεχτούν και ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο ότι δηλαδή ε, θα πρέπει ε, τουλάχιστον για τα οικονομικά στοιχεία η αναφορά να γίνεται αναέτος. Εγώ ε, θα ήθελα να ακολουθήσουμε την πρόταση του Επιτρόπου Μπαρνιέ και να εφαρμόσουμε και εδώ το ίδιο ζήτημα. Βεβαίως δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα αλλά σχετίζεται με το κείμενο το οποίο συζητήσαμε και εγκρίναμε πριν από μερικούς μήνες μήνες. Εάν δεν το κάνουμε τώρα δεν θα γίνει ποτέ ή θα αργήσει πάρα πολύ. Ε, και ε, ελπίζω, όπως είπαμε άλλωστε και για τις τηλεπικοινωνίες, ότι έχουμε μπροστά μας εκλογές. Ε, ας δράξουμε λοιπόν την ευκαιρία της ε, κίνησης που δημιουργείται λόγω των ε, εκλογών ε, και επομένως να πάρουμε αποφάσεις. Ναι, συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να υπερφορτώσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά να μην αφήσουμε να ξεγλιστρήσουν εύκολα και οι μεγάλες εταιρείες γιατί νομίζω ότι εάν και εμείς είμαστε σωστοί τότε και οι ανταγωνιστές μας θα είναι σωστοί. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας είπατε. Ο Σέλβος ο τελευταίος συγγεγραμμένος και μετά θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπέντσεν ε, για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνει για αυτά τα τόσο τεχνικά ζητήματα. Θα ήθελα να υποβάλω κι εγώ μία ιδέα, δεν ξέρω αν θα τη δεχτεί ε, ε, με αυτή την αναθεώρηση ενισχύουμε την ε, κοινωνική διάσταση. Λέμε ότι ε, δίνονται πληροφορίες κοινωνικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των μη χρηματοπιστωτικών πληροφοριών. Πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτές τις λογιστικές οδηγίες όπως και άλλα νομοθετήματα ώστε να μπορέσουμε να εισαγάγουμε και μία δεύτερη υποχρέωση για τις φορολογικές πληροφορίες εφόσον ε, πρόκειται για τη λογιστική οδηγία, διότι για τους διεθνείς ομίλους ε, τι θα ζητάμε ουσιαστικά, θα τους ζητάμε να δημοσιεύσουν κατάσταση ε, φόρων που έχουν καταβάλει στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί το λέω αυτό, διότι βλέπουμε από τις εργασίες της ομάδας G20 ότι υπάρχουν παράνομες δραστηριότητες, παράνομα κέρδη ε, και μεταφορά κερδών ανάμεσα στις θηγατρικές ενός ή δύο μήλου. Ε, γι' αυτό ξαναδιάβασα την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τιμολόγηση των υπηρεσιών που μεταφέρονται από τη μία θηγατρική στην άλλη. Δεν μπορούμε να ε, υποχρεώσουμε τους ομίλους με ένα συγκεκριμένο φορολογικό μορφότυπο να δηλώνουν πόσους φορούς ε, πληρώνουν στη χώρα όπου παράγουν. Η Google καλό θα ήταν να μας πει πόσους φορούς πληρώνει στην Αυστρία και στη Γερμανία κατά αναλογία με τις δραστηριότητες που έχει στην επικράτεια αυτών των χωρών. Όχι ότι θα το λύσουμε το πρόβλημα, αλλά θα έχουμε ένα πρώτο στοιχείο που εξασφαλίζει μια μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο εισηγητής, αλλά ε, καλό θα ήταν κατά τη γνώμη να προβληματιστούμε γι' αυτό. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή για να απαντήσει, θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Μπερνιέ Αμπάντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για τα σχόλια όλους τους ευρωβουλευτές. Τον Απρίλιο η Κομισιόν υιοθέτησε μια οδηγία που είναι συμβιβαστική λύση επιτρέπει στις βιομηχανίες μας να είναι σε ηγετική θέση στον τομέα αυτό αλλά προσπαθεί επίσης να αποφύγει υπερβολικό βάρος για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες. Στόχος μας, με βάση και τις μελέτες που κάναμε, είναι οι επιχειρήσεις όταν ε, σχεδιάζουν τη στρατηγική τους και τις συνεργασίες τους να εξετάζουν όχι μόνο τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και τις επιπτώσεις της, δραστηριότητάς τους, της δραστηριότητάς τους στο περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες κτλ. Αυτές οι επιχειρήσεις που το κάνουν αυτό είναι οι πιο επιτυχημένες μακροπρόθεσμα και οικονομικά και γενικότερα. Και έχουμε αρκετά στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η νομοθεσία αυτή είναι υπέρ των επιχειρήσεων. Αυτό μας λένε και οι επενδυτές. Ότι χρειάζονται αυτή την πληροφόρηση για να μπορούν να αντιμετωπίσουν ε, πλήρως πώς εξελίσσονται οι εταιρείες, πώς θα αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις κτλ τονίζουν ότι δεν υπάρχει αρκετή περιβαλλοντική και κοινωνική πληροφόρηση από τις εταιρείες που να επιτρέπει όλοι να εξετάζουν την πληροφόρηση αυτή. Εμείς ως Ευρώπη είμαστε στην πρώτη θέση. Είμαστε στην πρωτοπορία της ε, προσπάθειας αυτής. Λίγες χιλιάδες επιχειρήσεις ε, αναφέρουν όλα αυτά τα στοιχεία, είναι εντελώς διαφανής. Θέλουμε να αυξηθεί αυτός ο αριθμός, να περάσουμε στις 18.000 μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 500 εργαζόμενους στην Ευρώπη. Να είναι σαφές δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να χορηγούν αυτή την πληροφόρηση. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που έχουν ε, στην Ευρώπη πάνω από 500 εργαζόμενους θεωρούμε ότι είναι, υπολογίζουμε ότι είναι περίπου 18.000 και εκεί λέμε ότι στις ε, εκθέσεις της ε, διαχείρισής τους ε, καθώς ε, παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία. Πρέπει να παρουσιάσουν και αυτά τα στοιχεία, ώστε όλοι οι αναλυτές, οι επενδυτές κτλ. να έχουν μια πλήρη εικόνα. Να έχουμε λοιπόν στοιχεία για την επίπτωση της δράσης τους στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην απασχόληση, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άκουσα τα σχόλια και όλα τα θέματα της αλυσίδας προμηθευτών. Βεβαίως έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, διαφθορά και δωροδοκίες. Και επίσης στοιχεία και για τις ε, αμοιβέ των ε, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνον. Είναι λοιπόν νομίζουμε ισορροπημένη η πρότασή μας, αναφερόμαστε όχι μόνο στο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια, γιατί θέλουμε να αναγνωρίσουμε την αξία ορισμένων εθνικών προδιαγραφών για τις ορισμένα κράτη-μέλη, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, υπάρχει ο κανόνας βιωσιμότητας εκεί και η γαλλική νομοθεσία περιλαμβάνει πολύ σκόπιμες ε, διατάξεις που μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την παροχή πληροφοριών. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα εθνικών νομοθεσιών που συμπληρώνουν τις διεθνείς προδιαγραφές αναφέρθηκε ήδη ε, ο Σάκη, καθευτήρες γραμμές του, αλλά και η σφαιρική πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων και οι κατευθυντήρες γραμμές για ανθρώπινα δικαιώματα των ΗΕ. Υπάρχουν μια σειρά, μια σειρά σημεία αναφοράς. Ε, η, παγκόσμια μάχη των ΗΕ, όπως λέγεται, και αναγνωρίζουμε λοιπόν και τις εθνικές προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα ξαναδώσω τον λόγο σας, Αφρο Μπέντσιν για, για τα συμπεράσματά του. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ε, σκιώδεις ε, για τη συνεισφορά τους. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να τονίσουμε πως όταν συζητούμε για μια πιθανή εξαίρεση για τις μικρομεσαίες, όπως βλέπουμε σε κάποιες τροπολογίες, θα λέγαμε ότι ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε. Στη χώρα μου, παραδείγματο, χάρη από την εμπειρία μου, θεωρώ ότι ε, οι επιχειρήσει οι ίδιε θα πρέπει να διαβλέπουν τα ωφέλη του να συμμετέχουν σε μια στρατηγική εταιρική κοινωνική ευθύνη για να λειτουργήσει το σύστημα. Στη Δανία ισχύει η αρχή της ε, συμμόρφωσης ή αιτιολόγησης για μη, της Μετά από κάποια χρόνια εφαρμογής της αρχής βλέπουμε ότι το 97% των μεγάλων εταιριών ακολουθούν μια τέτοια στρατηγική ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δεν είναι ότι υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις να μας προσκομίζουν ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, τυποποιημένων πληροφοριών και όντως αληθεύει ότι αυτό ε, συνεπάγεται κάποια γραφειοκρατία. Όμως πρέπει να απαντηθούν ε, κάποια ερωτήματα, συγγνώμη, ούτως ώστε να δείξει η επιχείρηση ποια είναι η προστιθέμενη της αξία. Δεν είναι μια άσκηση όπου του ζητάμε να συμπληρώσουν κάποια πεδία ε, σε απλές ερωτήσεις. Πρόκειται για την κοινοποίηση των δραστηριοτήτων ε, της επιχείρησης. Αν δείτε την εμπειρία σε χώρα όπου ισχύει αυτή η αρχή και εφαρμόζεται αυτή η πολιτική εδώ και χρόνια θα συνειδητοποιήσετε ότι έχει νόημα και για τις ίδιες επιχειρήσεις ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις πληροφορίες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Σας διαβεβαιώ ότι στη Δανία, στη χώρα μου, ε, οι, οι απαιτήσει που υπάρχουν για την προσκόμιση πληροφοριών από πλευρά των επιχειρήσεων ε, έχουν κάποια συγκεκριμένη ωφέλεια. Ε, μιλώντας για την τις απόψεις των συναδέλφων θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω και σίγουρα απέφχομαι κι εγώ την αύξηση της γραφειοκρατίας. Ε, αλλά δεν, ε, το θέμα μας δεν είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Να ευχαριστήσω επίσης και τον Ζαν Πιερ και θα συζητήσουμε τη νέα ιδέα που κατέθεσε. Ευχαριστώ. Ωραία, υπενθυμίζω ότι 3 Οκτωβρίου εκπίπτει η προθεσμία ε, για την υποβολή τροπολογιών και η ψηφοφορία θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου. Έχουμε λοιπόν ακόμα μια εβδομάδα. Ε, ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο, ευχαριστούμε και όσους παρενέβησαν. Περνάμε στο επόμενο σημείο γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση αξιολόγησης ε, του Μπέρεκ. Θα δώσω αμέσως ε, τον λόγο ε, στον εισηγητή Σεντόι Ιαλαμπάρτ. 15-20 λεπτάκια έχουμε για αυτό το σημείο της μερισίας διατάξεως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν άμεσα τη συζήτηση. Τον εισηγητή παρακαλώ να παρέμβει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος όσον αφορά την έκθεση αυτή για τον Μπέρεκ ε, και την ε, αξιολόγηση του Μπέρεκ και τις ε, υπηρεσίες. Στόχος αυτής της έκθεσης είναι να κάνει μια πρώτη αξιολόγηση του φορέα για όσους δεν γνωρίζουν τον Μπέρεκ, πρόκειται για τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις ηλεκτρονικές ε, επικοινωνίες. Δηλαδή προσπαθεί να ρυθμίσει την αγορά των τηλεπικοινωνιών <clears throat> στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργήθηκε το 2009 με τη δέσμη τηλεπικοινωνιών Telecom. Ε, και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την πάροδο κάποιων ετών λοιπόν, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέω να κάνει μία έκθεση αξιολόγηση επί της οποίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει γνώμη. Ε, αυτός είναι και ο στόχος λοιπόν του της εδώ της γνωμοδότησης. Σε γενικές γραμμές το Μπέρεκ λειτουργεί καλά. Ε, φαίνεται να έχει δώσει την δυνατότητα ε, περαιτέρω ενδυνάμωσης της αμοιβαία εμπιστοσύνης και να έχει συμβάλει επομένως την επίτευξη των στόχων που εξ αρχής είχαν τεθεί. Ε, βεβαίως ε, υπάρχει δυνατότητα για ε, μεγαλύτερη, για περισσότερο φιλόδοξη εσωτερική αγορά ε, και το Μπέρεκ θα πρέπει να προετοιμαστεί γι' αυτό. Ε, το Μπέρεκ και η υπηρεσία πρέπει να είναι σε... Ε, έχουν και κάποια προβλήματα. Από την μία πλευρά βεβαίως αναγνωρίζεται η αξία της εργασίας του Μπέρεκ και της υπηρεσίας από τη δημιουργία του το 2009 κυρίως όσον αφορά το αρθρο 7 και 7α, τη διαδικασία δηλαδή των άρθρων 7 και 7α όσον αφορά την διεθνή περιαγωγή. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης, ε, κυρίως όσον αφορά κάποια ε, στοιχεία τα οποία αφορούν τις διεθνείς επικοινωνίες και που θα πρέπει να, να θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν, να τροποποιηθούν. Σύμφωνα με την αξιολόγηση, ο ανεξάρτητος λόγος ε, της ε, Μπέρεκ ε, δεν είναι απόλυτος και επομένως ακόμα τίθεται υπό αμφισβήτηση και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λογοδοσίας και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Επίσης ο ρόλος του Μπέρεκ θα πρέπει περαιτέρω και καλύτερα μάλλον να αποσαφινιστεί. Από ποιον προς ποιον λοιπά. Τέλος, ε, ο τόπος εγκατάστασης στην, της Μπέρεκ, στη Ρήγα δηλαδή, ενδεχομένως είναι ε, δύσκολο να παρακολουθεί την ε, διαρκώς εξελισσόμενη κατάσταση. Δύο βασικές προσεγγίσεις μπορούν να τεθούν προς εξέταση για το σχέδιο έκθεσης. Μία στατική προσέγγιση η οποία μπορεί να, είναι, να, να πει ότι η τρέχουσα είναι σαφώ καθορισμένη και επιτυχή και δεν απαιτούν σημαντικέ αλλαγέ, αλλά και μια εξελικτική προσέγγιση. Δηλαδή να θεωρήσουμε ότι είναι επιτυχή μεν η υπάρχουσα δομή, αλλά ότι μπορεί να προσδιοριστεί καλύτερα ε, και ότι επομένω θα πρέπει μια πιθανή λύση να είναι η παραχώρηση περισσότερων αρμοδιοτήτων και εγκατάσταση του Μπέρεκ ε, στι Βρυξέλλε. Άλλωστε υπάρχει εδρεωμένη παρουσία της, ε, του, του Μπέρεκ. Η αξιολόγηση ε, όσον αφορά την υπηρεσία καταδεικνύει ότι είναι ακόμα αμφιλεγόμενη ε, η θέση της ε, υπηρεσίας και όσον αφορά την δική του λειτουργία και όσον αφορά την λειτουργία του σε σχέση με τον κανονισμό Μπέρεκ. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσουμε με την Κατρίν ε, Τρότμαν. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με τους ε, σκιώδεις. Η κυρία Τρότμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε στην αρχή είχε προταθεί από την Επιτροπή μια υπηρεσία που θα ονομαζόταν ΕΚΜΑ ε, και που δεν έγινε δεκτή και από τα κράτη-μέλη και από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Ε, επελέγει μια υβριδική μορφή έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ε, να υλοποιηθεί καλύτερα και να υλοποιηθεί καλύτερα το πλαίσιο. Η ιδέα ήταν ε, σιγά σιγά ε, οι ρυθμιστικές προσεγγίσεις ε, να συγκλίνουν κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία του άρθρου 7 και 7α. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή γιατί πολύ ορθά αντιμετώπισε το ζήτημα και ορθώς επίσης κάνει προτάσεις όσον αφορά τα σημεία τα οποία παραμένουν ακόμα εκκρεμή ενώ διαπιστώνει ότι υπάρχουν και θέματα στα οποία τον Μπέρεκ έχει ε, ε, προχωρήσει σωστά. Τα κυριότερα προβλήματα τα οποία υπογραμμίζονται είναι πρώτα ο τόπος εγκατάστασης. Τόπος εγκατάστασης που άλλωστε δεν αφορά μονάχα αυτή την υπηρεσία και αυτό το φορέα. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να αντισταθούμε ε, στην, ε, στην πρόκληση αυτή που έχουμε για επικέντρωση των υπηρεσιών ή διαφορετικά θα πρέπει ειλικρινά να πούμε στις περιφερειακές χώρες πιο απομακρυσμένες ότι δεν θα μπορούν να έχουν καμία παρουσία στο έδαφος τους οποιοδήποτε φορέα. Όσον αφορά τώρα το ε, πεδίο ε, ε, της λειτουργίας του Μπέρεκ. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα έλλειψης ομοιογένειας μεταξύ των εθνικών εθνιστικών αρχών και όσον αφορά τις δικαιοδοσίες τους και άλλωστε αυτό αναφέρεται και από τον εισηγητή στο σημείο 6. Εκεί λέει ο εισηγητής ότι το το πεδίο, το, η δυνατότητα μάλλον ε, ε, ελιγμών που έχουν οι χώρες είναι πάρα πολύ μικρό. Επίσης, η δυναμική σε σχέση ανάμεσα στο Μπέρεκ και την υπηρεσία. Τι να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει, να διαλυθεί η υπηρεσία. Αλλά αυτή είναι μια επιλογή ε, του ε, ε, Συμβουλίου που δεν είχε γίνει δεχτή. Αυτό θα σήμαινε ταυτόχρονα ότι οι εθνικές διεθνικές αρχές θα έπαιρναν πάρα πολύ μεγάλο βάρος και επομένως ε, θα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο. Ε, πιστεύουμε ότι και από την άποψη της ε, ανεξαρτησίας όλου του τομέα καλό θα ήταν να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στον φορέα και την υπηρεσία έτσι ώστε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία αφενός αλλά αφετέρου να υπάρχει και η δυνατότητα αποφάσεων από πλευράς του φορέα Ωραία. Ε, τώρα θα μπορούσαμε ε, να δούμε το ενδεχόμενο ε, να έχει η υπηρεσία δικούς τις πραγματογνώμονες που θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο άρθρο 7 και 7α αλλά να έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά μετά από πρωτοβουλία του Μπέρεκ. Αυτά σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Κατρίν Τροτμάν. Δεν έχουμε άλλους σκιώδεις παρόντες. Επομένως δίνω το λόγο στην Πλήρα Δεκαστήλιο. Ε, Ευχαριστώ. Συγχαίρω τον εισηγητή για την πρόταση που μας κάνει για να εκτιμήσουμε το Μπέρεκ. Χαίρομαι πολύ που συζητάω τον Μπέρεκ γιατί ήμουν εισηγήτρια για τον Μπέρεκ όταν ζητήσαμε το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες, το Μπέρεκ ε, προέκυψε ως μια εναλλακτική λύση στην πρόταση δημιουργίας ε, ενός οργανισμού, ευρωπαϊκού οργανισμού με όλη τη δομή που έχουν αυτές οι, αυτοί οι οργανισμοί. Έτσι πρότεινε τότε η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, όπως και το Συμβούλιο, ε, προτίμησε την αναλλακτική λύση να δημιουργηθεί αυτός ο φορέας με βάση τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Οπότε το Μπέρεκ είναι πρόσφατη εξέλιξη. Τρία χρόνια λειτουργεί. Και όπως λέει και ο συγητής, ανέφερε πόσο θεμελιώδες είναι το άρθρο 7, πόσο σημαντική είναι η επιτήρηση της ουδετερότητας του διαδικτύου. Δεν νομίζω ότι το Μπέρεκ θα έπρεπε να αναθεωρηθεί ριζικά από πλευράς δομής, αλλά η προσέγγιση του εισηγητή, όπως την εξήγησε και η κυρία Τρότμαν, πρέπει κάπως να διευκρινιστεί περαιτέρω, να εκλεπτυνθεί. Συνδέοντας τη συζήτηση με την προηγούμενη, που είχαμε με την Επιτροπή για την πρόταση κανονισμού για την εσωτερική αγορά τηλεπικοινωνιών όπου γίνονται πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τον Μπέρεκ. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον και θα ε, προκαλούσε θετικές, ε, θετικά, θρηστικά αποτελέσματα αν συνδυάζαμε τα δύο αυτά θέματα. Να εξετάσουμε δηλαδή κάποιες προτάσεις που κάνει η Επιτροπή. Μία νομίζω ότι είναι σημαντική. Και άλλες μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά μία που είναι και εύκολα κατανοητή αυτή η δυνατότητα το Μπέρεκ να έχει πρόεδρο για μεγαλύτερη θητεία. Τώρα γίνεται κάποια εναλλαγή κάθε 6 μήνες. και συμφωνώ με αυτό που είπε πρόσφατα η Επίτροπος ότι είναι πολύ μικρό αυτό το διάστημα της θητείας. Γίνονται συνέχεια αλλαγές. Αυτό δεν είναι καλό για την ε, συνέπεια της δράσης του Μπέρεκ και τη συνέχεια. Θα ήταν σκόπιμο λοιπόν, μια που συζητάμε τον απολογισμό του Μπέρεκ, δεν είναι νομοθετικό θέμα, να εξετάσουμε και αυτή την πρόταση αλλά και άλλες. Γιατί κάποιες θα μπορούσαν ήδη να συμπεριληφθούν στη διαδικασία τροπολογιών. Ευχαριστώ και εκ νέου τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Η δόκτωρ Νικολίτα Φαλκόνη έχει το λόγο, εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα δώσουμε ξανά το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την έκθεση, την οποία με μεγάλη προσοχή παρακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, χαιρόμαστε γιατί ορισμένα από τα συμπεράσματα στα οποία είχε καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάρκεια της αξιολόγησης ε, αναφέρονται στην έκθεση εδώ από τον εισηγητή. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια ε, στοιχεία που που ακολουθούν τελικά την ίδια γραμμή των συμπερασμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκθεση αξιολόγησής της. Επομένως, ε, η δικιά μας γραμμή είναι ότι το Μπέρεκ λειτουργεί καλά, ότι απέδειξε ότι έχει την δυνατότητα να καλύψει τον ε, θεμελιώδη στόχο δηλαδή τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς, αλλά ταυτοχρόνως έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία χρήζουν βελτιώσεως. Ε, θα ήθελα κυρίως να λάβω υπόψη μου και την ε, παρέμβαση που έκανε η κυρία Καστίγιο και εμείς ε, θεωρούμε ότι το Μπέρεκ θα πρέπει να βελτιώσει την στρατηγική του θέση. Ε, πρέπει όμως ε, να ε, να υπάρχει και μεγαλύτερη σταθερότητα στην διακυβέρνηση της ε, υπηρεσίας. Ε, γι' αυτό έχει κάνει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η οποία έγινε δεκτή πρότεινε να υπάρξει στα πλαίσια του Μπέρεκ μια νέα θέση, η θέση του Προέδρου, έτσι ώστε να μην υπάρξει αυτή η ε, εναλλαγή στην Προεδρία, να υπάρχει καλύτερη δυνατότητα ε, διαχείρισης ε, της Μπέρεκ και ταυτοχρόνως να υπάρχει δυνατότητα στρατηγικής σταθερής ηγεσίας. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε τον λόγο τώρα ξανά στον, λόγο, τον συνάδελφο Σεντόγια Αλαμπάρτ. Ευχαριστούμε Πρόεδρε. Να πω ότι είχα από πλευράς ε, ε, της ε, πολιτικής ομάδας και των άλλων πολιτικών ομάδων την θέση τους η ε, συνάδελφη από του πράσινου μου την έστειλε άλλωστε γιατί δεν ήταν εδώ. Εν πάση περιπτώσει θα αναλύσουμε τι ε, τροπολογίε. Ε, θα δούμε ποια είναι η ανάλυση που μπορούμε να κάνουμε των προσεγγίσεών του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την πληρέστερη αξιολόγηση του Μπέρακ και τη Υπηρεσία. Ευχαριστώ πολύ. 2 Οκτωβρίου η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, ψηφοφορία στι 5 Νοεμβρίου. Επόμενο σημείο ε, είναι ένα θέμα ακανθόδες, να το πούμε έτσι. Κατεξουσιοδότηση κανονισμός ε, για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης στο GEMS οι Στέφη Κρότσμαν, ε, ε, ε, Μπράουξ και Ιντάρ έχουν υποβάλει ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εκεί ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Θα δώσω πρώτα απ' όλα τον λόγο στον κύριο Κρότσμαν. Ξέρετε ότι η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Παρακαλώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι ως ένας από συνυπογράφουν ε, το ψήφισμα για αυτήν την εξορλουσιοδημένη πράξη, να σας πω τα εξή Με αυτή την πράξη, ε, μετά από τρία χρόνια, προτείνει την εφαρμογή του κανονισμού GMES. Ε, θα παίρνονται έτσι οι κεντρικές αποφάσεις. Άρα η διάθεση χωρίς τελική, χωρίς, ε, ε, χωρίς ε, αμοιβή όλων των στοιχείων που συλλέγει το σύστημα Sentinel. Σε μια συνάντηση με την Κομισιόν μας διευκρινίστηκε ότι λόγω των της διαφορετικής, ε, διαφορετικού επίπεδου λειτουργίας των συστημάτων δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού αλλά οι επιπτώσεις δεν έχουν αναλυθεί κατά τη γνώμη μου ε, ε, δεν έχει γίνει σωστή ανάλυση. Θα δίνουμε και στους Αμερικανούς αυτά τα στοιχεία χωρίς κόστος. Όμως το σύστημά τους έχει εντελώς διαφορετική ανάλυση. Και γι' αυτό ακριβώς η σύγκριση δεν ισχύει. Και δεν είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι δεν έχει κόστος αυτό, διότι τους ε, δορυφόρους αυτούς τους πληρώνει ο Ευρωπαίος φορολογούμενος. Βεβαίως, μέσω της χρήσης θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Όμως, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα δίνουμε σε όλους δωρεάν αυτά τα στοιχεία. Μόνο ορισμένα στοιχεία, ορισμένα είδη στοιχείων ή παλαιότερα στοιχεία θα μπορούσε να είναι ελεύθερα προσβάσιμα. με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια αγορά στους ιδιωτικούς επενδυτές που έχουν ήδη κάνει σημαντικές επενδύσεις. Τώρα και τρίτα κράτη θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση ενώ δεν έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση. Κατά τη συζήτηση για τον κανονισμό το συζητήσαμε αυτό και είχαμε πει ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια αρχή αμοιβαιότητας. Το σύστημα GMES δεν είναι ότι δίνει δωρεάν τα στοιχεία, δεν είναι αυτό το πλεονέκτημά του. Αλλά το θέμα είναι, ποια είναι ποιες είναι οι συνθήκες. Ένα σημαντικό θέμα πρέπει να το λύσει ο νομοθέτης. Και όχι μέσω κατεξοδότηση πράξης. Η Επιτροπή μοιάζει να το αναγνώρισε αυτό, γιατί ο νέος κανονισμός ε, για τον Κοπέρνικο το προβλέπει, Κοπέρνικος το προβλέπει συγκεκριμένα. Τώρα δεν είναι σαφές επίσης αν αυτή η κατεξοδότηση πράξη θα βασίζεται στον παλιό κανονισμό. Θα μπορούσαμε να περιμένουμε γιατί είναι σημαντικές οι αποφάσεις που θα λάβουμε. Έχουμε περιμένει τρία χρόνια, μπορούμε να περιμένουμε μερικούς μήνες ακόμη. Για αυτούς τους λόγους που είναι περιεχομένου και ε, διαδικαστικούς σας προτείνω να απορρίψουμε αυτήν την κατεξοδότηση πράξη, ούτως ώστε η απόφαση να πάρθει με βάση το νέο κανονισμό για το Κοπέρνικο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ στον άλλον υπογράφοντα ε, του, του ψηφίσματος, ο κύριο Γκλάντ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ψήφισμα και οι συγητές ε, προκάλεσαν κάποια σύγχυση. Και στη δική μου ομάδα, αρχικά περί σε επρόκειτο, στα πλαίσια του κανονισμού GMES, όπου είχα εργαστεί και εγώ, να ρυθμίσουμε ε, την πρόσβαση στα στοιχεία και ότι θα ήταν δωρεάν. Αλλά δεν τα είχαμε ρυθμίσει ε, αρκετά σαφώς και γι' αυτό χρειάζεται τώρα εξοδότηση πράξη. Πήραμε αυτή την πρόταση λίγο πριν τις διακοπές για την κατεξοδότηση πράξη και είχαμε μέσω των αγκαίων υπογραμμών, υπογραφών ζητήσει να ε, παραταθεί προθεσμία τόσο ώστε αυτή η νέα κατοριστότηση πράξη να λεφθεί με βάση τον νέο κανονισμό. Η ομάδα μου το εξέτασε αυτό και με βάση αυτά που είπε ο Σάνθος Κρότσμαν θεωρούμε ότι εφόσον έχει υποβληθεί ο νέος κανονισμός να τον συζητήσουμε και ο κανονισμός 15 του νέου κανονισμού αναφέρεται στην ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση και αποφασίσαμε να απορρίψουμε το ψήφισμα για να μην υπάρξει πενταρό καθυστέρηση. Ήδη έχουμε καθυστερήσει αρκετά και συζητήσαμε και το θέμα της μελλοντική χρηματοδότηση του Κοπέρνικου. Είμαστε υπέρ λοιπόν να εγκριθεί αυτή η κατεξοδότηση πράξη και να επικεντρωθούμε σε αυτόν τον νέο κανονισμό Κοπέρνικος, τον οποίο θα συζητήσουμε αναλυτικά. Νομίζω ότι αυτή είναι ε, λογική λύση και θα συμφωνήσουν επ' αυτού οι ομάδες αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Σούλτεμπραξ, αν δεν κάνω λάθος. Γεια σας, είμαι επικεφαλής τμήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις υποδομές ε, Κοπέρνικους και για τα θέματα πρόσβασης ε, στα δεδομένα στους τομείς αρμοδιότητας της μονάδας μου. Σημείωσα ότι το σχέδιο ψηφίσματος αναφέρεται σε τυπικά ζητήματα. Έχει σημειωθεί καθυστέρηση, δηλαδή μπορούμε να αναβάλουμε το ζήτημα για λίγους μήνες, όμως δεν υπάρχει αναφορά στο περιεχόμενο, στην ουσία. Εμείς αυτό θα προτιμούσαμε, να γινόταν σήμερα μια συζήτηση για την ουσία. Είμαι ε, ο πρώτος που λυπάται για την καθυστέρηση. Πριν από ένα χρόνο ανέλαβα τα καθήκοντά μου μόλις. Είχε, είχαν γίνει προπαρασκευαστικές εργασίες, διαβουλευτήκαμε με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς επανειλημμένα. Προετοιμάσαμε διάφορες εκδοχές του κειμένου, διαδοχικές εκδοχές, τις οποίες αποστήλαμε ε, για σχολιασμό στους εμπλεκόμενους φορείς. Δεν γίνεται σπευσμένα να ε, καταθέσετε μία πρόταση ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται και την συνενετική άποψη των εμπλεκομένων ε, φορέων. Εμείς ε, επιδιώξαμε το δεύτερο κατά προτεραιότητα και το πετύχαμε. Και μας ξάφνιασε ότι μόνο μία εταιρεία η οποία τώρα κάνει ασκεί ειδική πίεση στο, στο κοινοβούλιο δεν συμφώνησε. Ε, διότι οι δορυφόροι της ε, ανταγωνίζονται ε, τους δορυφόρους της πρωτοβουλίας Sentinel-2. Αυτό το ξέραμε όμως χρόνια τώρα και το, έχουμε συζητήσει με το είχαμε τότε συζητήσει επανειλημμένα με την γερμανική κυβέρνηση και λήφθη η απόφαση το Sentinel-2 να απορρίψει έναν αισθητήρα που ε, συνιστά επικάλυψη με τα ε, συστήματα ε, των δορυφόρων αυτής της εταιρεία. Η ανάλυση είναι 500 μέτρα και ξεπερνάει τη δική μας ανάλυση κατά 400%. Οπότε αφήσαμε περιθώριο ελιγμών σε αυτή την εταιρεία και αποστασιοποιηθήκαμε. Φαίνεται ότι τώρα έχει ξεχαστεί αυτό. Ήταν τεράστια παραχώρηση από πλευράς μας. Η εταιρεία επένδυσε σε αυτούς τους δορυφόρους παρότι γνώριζε την κατάσταση. Αυτή είναι, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και ο αισθητήρα τους πάλι υπερβαίνει σε απόδοση τους δικούς μας, τουλάχιστον κατά 1000%. Παρόλα αυτά μπορούν να έχουν ε, εφάμιλες εμπορικές δραστηριότητες. Κάτι άλλο που τους ενοχλεί είναι το εξής θα έχουμε σταθερές ε, συνθήκες, συνθήκες πλαίσιο μελλοντικά. Ναι. Είναι καταφατική απάντηση, διότι το μακροπρόθεσμο σενάριό μας προβλέπει ότι η ανάλυση των δορυφόρων μας δεν θα αναβαθμιστεί για τα επόμενα χρόνια και αυτό μέχρι το 2026. Η εταιρεία αυτή που κάνει το lobbying έχει σταθερές επιχειρησιακό περιβάλλον για τα επόμενα 13 χρόνια. Λίγες εταιρείες μπορούν να πούν ακριβώς το ίδιο. 13 χρόνια. Είναι ο κύκλος ζωής δύο γενιών δορυφόρων. Κάθε γενιά κρατάει, έχει κύκλο ζωής ε, μία εφταετία. Μπορούν λοιπόν να επενδύσουν ε, κατά τη διάρκεια αυτή τη περίοδου δεν θα αυξηθεί ο ανταγωνισμό από πλευρά των δορυφόρων Sentinel-2. Και δεν καταλαβαίνουμε γιατί προτείνεται απόρριψη. Ε, Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να πάρετε το λόγο, Σνάλφε Κρότσμαν. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν θέλω να σχολιάσω. Αύριο θα ψηφίσουμε. Ε, επειδή φεύγατε, ήθελα να σας σταματήσω για αυτό μόνο, αν θέλατε να πάρετε το λόγο πριν φύγετε. Ο κύριος Οντή. Ε, ομολογώ ότι είναι λίγο μυστηριώδης αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Μάλλον δεν έχω αρκετή εμπειρία και δεν καταλαβαίνω. Ίσως δεν τα κατάλαβα όλα ή δεν τα διάβασα όλα, αλλά εγώ από ό,τι θυμάμαι για το GMES μιλήσαμε και για τιμολόγηση. Εγώ ήμουν υπέρ και συμφωνήσαμε όλοι ότι πρέπει να είναι δωρεάν η διάθεση. Και δεν καταλαβαίνω εξάλλου γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται νομική βάση για τη δωρεάν διάθεση στο μέτρο που αυτό καλύπτεται από την αρχική νομική βάση. Για ποιο λόγο χρειάζεται αυτός ο κανονισμός. Τώρα μαθαίνουμε ότι πλήττεται μια ιδιωτική εταιρεία λόγω των δημοσίων επενδύσεων, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν όρια στη δημόσια παρέμβαση και ποια είναι αυτά, όταν καταρρεύσει και εκλείψει η ιδιωτική πρωτοβουλία, για ποιο λόγο δεν μπορούμε να παρέμβουμε δημοσίως. Και τώρα Υπάρχει εμπλοκή για το πρόγραμμα GMS e και έχουν ενημερωθεί στο μεταξύ ε, οι πολίτε ε, για την προστιθέμενη αξία, για τους πάγους που λιώνουν και μπλα μπλα μπλα και μπλα μπλα μπλα. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται νέα νομική βάση για δωρεάν διάθεση πληροφοριών εφόσον το έχουμε ήδη εγκρίνει διαψήφου και ε, γιατί αυτή η εταιρεία ακόμη εξακολουθεί να κάνει λόμπινγκ για να καθυστερήσει αυτό το τόσο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ε, έχω θορυβηθεί, δεν το κρύβω. Πρόεδρος. Ωραία τα έχουμε ακούσει όλα, τα παρακολουθήσαμε όλα, επομένως ε, αύριο θα ε, ψηφίσουμε έτσι ώστε, μάλλον θα έχουμε τη δυνατότητα, αύριο αύριο στις 26 ε, Σεπτεμβρίου θα λάβει χώρα η ψηφοφορία, είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, τα έχουμε ακούσει όλα, ξέρουμε πολύ καλά με ποιο τρόπο θα ψηφίσουμε και η ψήφο στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο. Ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας, θα ξαναρχίσουμε στις 3 το απόγευμα.